ο κύριος πρόεδρος. Καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των υπερασπιστών των δασών και του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και πάλι ότι υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλετε έτοιμα για να σας δοθεί ο λόγος με τη διαδικασία του Catch the Eye και με τη διαδικασία της ερώτησης για τη γαλάζια κάρτα, χρησιμοποιώντας τόσο τη συνήθη διαδικασία, όσο και το ηλεκτρονικό σύστημα. Οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην είσοδο του ημικυκλίου. Εξ ονόματος της Επιτροπής, το λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Μίμητσα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω όλα τα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύσει και να αποκαταστήσει στην αρχική τους κατάσταση τα ευρωπαϊκά δάση αλλά και όχι μόνο. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, συνολικό θα έλεγα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά είναι τα δάση τα οποία προστατεύονται από την οδηγία Habitat, όπως επίσης και από την οδηγία για, τα προστατευόμενα ε, πτηνά. Στην παρούσα φάση το 23% των δασών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκει επίσης στο δίκτυο το λεγόμενο Natura 2000 με προστατευόμενα σημεία και υπάρχουν φυσικά και οι ε, οδηγίες που προστατεύουν συγκεκριμένα είδη ε, εμπειονόντων. Οι περασπιστές φυσικά του περιβάλλοντος είναι η φυσική μας σύμμαχοι για την προώθηση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Ένα άλλο μέσο είναι η οδηγία για τις ε, ποινικά κολάσιμες παρεμβάσεις στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να πάρει μέρος στον αγώνα εναντίον του εγκλήματος και διεξάγεται σε αυτή τη φάση και μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 μια διαβούλευση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας. Επίσης υπάρχουν και κανονισμοί σχετικά με τη δασοκομεία και τις ε, απαγορεύσεις σε περιοχές όπου ε, ε, υπάρχει ανάγκη έλεγχος. Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα είναι, θεωρούνται απειλή βάρος της ίδιας της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της ε, προσπάθειας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που έχει ξεκινήσει και διαρκεί μέχρι το 2021. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στις δυνάμεις ε, τις αστυνομικές, τις δυνάμεις καταστολής, έτσι ώστε να υπάρξουν λειτουργικές παρεμβάσεις προστασίας. Έχει σημασία να γνωρίζουμε εδώ ότι τα κράτη-μέλη είναι τα υπάρθυνα για την εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων, όπως επίσης και για την ε, λήψη μέτρων επιβολής, μεταξύ των οποίων πρόστιμα και κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των κανόνων και αναλαμβάνει δράση όποτε αυτό ε, απαιτείται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης παρέχει οικονομικούς πόρους για την αποκατάσταση αηφόρο διαχείριση ε, των δασών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ε, Στρατηγικής. Στα πλαίσια των ε, διαφθορτικών ταμείων και στα πλαίσια της κοινή αγροτικής πολιτικής υπάρχουν πόροι ε, οι οποίοι φτάνουν τα 8,2 δις στα πλαίσια της περίοδου 14-20. Τέλος, η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης για την προστασία και αποκατάσταση των δασών δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τις προσπάθειές της για την ε, προστασία της βιοπικιλότητας και την καταπολέμηση της απώλειας βιοπικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό πάλι θα πρέπει για μια ακόμη φορά να υπογραμμίσω τον σημαντικό ρόλο που έχει ε, η νομοθετική ρύθμιση ε, για τα προϊόντα τα δασικά είτε παράγονται στην Ένωση είτε εισάγονται από τρίτες χώρες. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στην παρούσα φάση ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις παράνομης δασοκομικής δραστηριότητας ακόμα και σε πρωτογενείς δασικές εκτάσεις ε, σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Για την ειδική περίπτωση της Ρουμανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για να αξιολογήσει την παρούσα κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης αναλύει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 μάλλον των γεωργικών εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλέπτονται από δασικές εκτάσεις. Αυτό δείχνει τη μεγάλη σημασία που έχουν οι δασικές εκτάσεις, ιδιαίτερα για περιοχές οι οποίες δεν έχουν πυκνή κατοίκηση. Σήμερα όλοι προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε ένα φαινόμενο χωρίς σύνορα, δηλαδή τις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών συνεπώς θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ε, σε επίπεδο πολιτικό όχι μόνο για την προστασία των υπαρχουσών δασικών εκτάσεων αλλά και για την ε, σωστή συντήρηση και αποκατάσταση των περιοχών που έχουν βλαφθεί Ευχαριστώ για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Το λόγο έχει η κυρία Αρένα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κάθε χρόνο οι άντρες και οι γυναίκες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος εκφοβίζονται. Πάνω από 160 άτομα έχασαν τη ζωή τους ε, γιατί υπεράσπισαν το περιβάλλον ε, το 2018. Και όταν δεν χάνουν τη ζωή τους, πολλές φορές συλλαμβάνονται ή τους απειλούν με χρήση βίας επειδή αντιτίθενται στις κυβερνήσεις και στα συμφέροντα των επιχειρήσεων που ουσιαστικά τους αρπάζουν ε, τις γέες και τα δάση τους. Αν η Ευρώπη δεν είναι αυτή η οποία πλήττεται περισσότερο. Δεν είναι και ε, προστατευμένοι από τέτοια φαινόμενα. Έχουμε παράνομη υλοτομία στη Ρουμανία. Στον Ηνωμένο Βασίλειο επίση καταδικάστηκαν τρία άτομα σε πολλά χρόνια ε, κράτηση λόγω παράνομων εξορρυκτικών δραστηριοτήτων ε, ε, σχιστολιθικού αερίου. Υπάρχουν παράνομε λοιπόν τέτοιε δραστηριότητε τι οποίε πρέπει να αντιμετωπίσουμε με δεσμευτική νομοθεσία ώστε οι εταιρείε να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους κατά των ακτιβιστών. Υπάρχει επίση αγωγή πρώτων υλών από τρίτε χώρες και θα πρέπει η Ένωση να φροντίσει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού σέβεται σήμερα ε, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Καλή νομοθεσία που έχουμε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο σε ό,τι αφορά την εταιρική ευθύνη. Οι ακτιβιστές του περιβάλλοντο ε, πρέπει να στραφούν στην Ευρώπη για να εξασφαλίσει την προστασία του όταν ε, είναι θύμα τέτοια βία δεν θα πρέπει να συγγύσουν ούτε να φημωθούν. Αυτοί οι ακτιβιστές αντίθετα να προστατευθούν και να τιμωρηθούν όσοι ε, καταστρέφουν το περιβάλλον. Ουσιαστικά αυτά τα φαινόμενα, αν δεν τα αντιμετωπίσουμε, κάνουμε έτσι να θεωρείται και ε, συνηθισμένο το φαινόμενο της ε, επίθεσης που δέχονται. Πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς και στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ για την ομάδα Renew Europe. Το λόγο έχει η κυρία Ροντρίγκε Ράμο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα δάση είναι η ζωή μας διότι φιλοξενούν το 30%, μάλλον καλύπτουν το 30% της επιφάνειας του πλανήτη μας, αλλά διατηρούν το 80% της βιοποικιλότητας. Χάρη στα δάση αναπνέουμε, ζούμε. Επομένως, με πολύ ικανοποίηση ε, σημειώνουμε την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των ευρωπαϊκών αλλά και παγκόσμιων δασών. Το σίγουρο είναι πως ε, όσο επιδεινώνονται οι συνθήκες ε, στα δάση, επιδεινώνονται επίσης οι συνθήκες διαβίωσης και δράσης των ακτιβιστών. Και έχουμε στοιχεία όπως το Frontline Defenders στην έκθεσή του το 2018 που λέει ότι 247 ηγέτες για περιβαλλοντικά ζητήματα, άνδρες και γυναίκες ε, είτε εγνοούνται είτε κακοποιήθηκαν είτε απειλήθηκαν γιατί προσπάθησαν ουσιαστικά να υπερασπιστούν ε, το φυσικό μας περιβάλλον, το δικαίωμα όλων μας στη ζωή. Η καταστροφή της βιοπικιλότητα όμως δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζετε μόνο με τη νομοθεσία. Θεωρείται και πρέπει να θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει μέτρα ώστε να υπερασπιστεί ε, όσους υπερασπίζονται το περιβάλλον μας. Πρέπει να βελτιωθεί η περιβαλλοντική νομοθεσία, να ρυθμιστούν καλύτερα τα περιβαλλοντικά δικήματα. Επίσης, έχουμε 40 οικολογικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίες διαμαρτύρονται, διαδηλώνουν και ζητούν δικαιοσύνη για την δολοφονία δύο δασοφυλάκων στη Ρουμανία, οι οποίοι κατα... κατήγγυλαν την παράνομη λοτόμηση. Το 43% του ξύλου από τα δάση στη Ρουμανία το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, προερχόταν από ε, πηγές οι οποίες ε, δεν έχουν πιστοποιηθεί. Θέλουμε λοιπόν ε, να μην υπάρχει απερίμωση των δασών ούτε στην Ευρώπη ούτε στη, στον κόσμο και πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προς αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το αναλάβει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Τούσαν. Ευχαριστώ. Οι δύο δασοφύλακες στη Ρουμανία έχασαν τη ζωή τους στο φθινόπωρο γιατί ήθελαν να προστατεύσουν τα δάση και πολλοί άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη μαφία των δασών στη Ρουμανία. Προστάτευαν το περιβάλλον. μας. κανείς όμως ε, δεν προστάτευσε αυτούς. Αυτούς που γίνονται στόχοι και το ξέρουμε κάθε χρόνο. Από 200 περασπιστές της φύσης χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. Κάθε εβδομάδα τρία άτομα χάνουν τη ζωή τους γιατί υπερασπίζονται ουσιαστικά τον πλανήτη μας απέναντι ε, στα συμφέροντα εξορρυκτικών ή ε, αγροδιατροφικών βιομηχανιών. Ε, δέχονται επιθέσεις, φημώνονται, τους συλλαμβάνουν, τους καταδικάζουν και Πολλέ φορέ του απειλούν και με θάνατο. Έχουμε λοιπόν την οικολογική, εγκληματική αυτή μαφία, αλλά και τα κράτη που με τις πολιτικές τους ουσιαστικά ποινικοποιούν και εκφοβίζουν τους ακτιβιστές. Ο κινησμό σκοτώνει, όπως και η ε, λεμαργία και η... είδαμε τι κάνει ο Μπολσονάρο, ο εμπορικός μα εταίρο. Σατζε Αλεγρία, τέσσερι ε, ε, υπερασπιστές του περιβάλλοντο κατηγορήθηκαν ε, αυτήν την εβδομάδα. Εκεί ήρθαν στο σπίτι τους ε, και έκαναν έφοδο και έψαξαν τα πάντα. Κρέμι Φρέσ. Με... Ε, έχασε τη ζωή του από πειρά τη γαλλική αστυνομία. Δεν είναι μόνο οι Ρουμάνοι, τα σοφύλακε, είναι πολλοί άλλοι. Με την ε, συνενοχή μα ε, δικαιολογούμε την συνέχιση τέτοιων φαινομένων. Πρέπει λοιπόν να πάψουμε να είμαστε συνένοχοι και θα πρέπει με αποφασιστικότητα και ισχύ να προστατεύσει η Ένωση αυτού που μα επιτρέπουν ακόμη και σήμερα να ζούμε σε ένα κατοικήσιμο πλανήτη. Για την ομάδα ταυτότητα και δημοκρατία, το λόγο έχει η κυρία Μπενιέ Συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεπεράσω το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι υπασπιστές του περιβάλλοντος είναι στόχοι στον κόσμο όλο. Σύμφωνα με Μίκιο 164 υπερασπιστές του περιβάλλοντος δολοφονήθηκαν πέρυσι εναντίον προγραμμάτων γεωργικών, δασικών, αγροβιομηχανικών και άλλοι αναγκάστηκαν να σιωπήσουν λόγω της βίας που ασκήθηκε εις βάρος τους. Είναι θλιβερή η κατάσταση. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Πρέπει φυσικά να πιέσουμε τα κράτη-μέλη που ενθαρρύνουν αυτού του είδους τα προγράμματα. Ε, πρέπει να βοηθήσουμε τους ηρωικούς υπερασπιστές του περιβάλλοντος αλλάζοντας και μορφές κατανάλωσης η παράνομη κυνηγητική δραστηριότητα υπάρχει διότι τα προϊόντα απολούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατανάλωση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 10% ε, των προϊόντων της αποψήλωσης των δασών στην Ιδρόγειο. Ε, είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να καταναλώνουμε από εδώ και πέρα με οικο-υπεύθυνο τρόπο και να σταματήσουμε τις πρακτικές λαιλασίας των δασικών πόρων. Ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, το λόγο έχει ο κύριος Σλαμπάκοφ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω την εντύπωση ότι χρειαζόμαστε νέου τύπου κανονισμούς για να υπερασπιστούμε το περιβάλλον. Νομίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν την κατάλληλη νομοθεσία προστασίας ε, των δασών τους. Και γιατί δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε και τους υπερασπιστές όπως λέγεται του περιβάλλοντος. Γιατί πολλές φορές ε, οι άνθρωποι αυτοί ε, σαμποτάρουν, υπονομεύουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και χρησιμοποιούν τις πιστώσεις της ευρωπαϊκές με καταχρηστικό τρόπο. Η οικολογία λόγω αυτών των ανθρώπων έχει μετατραπεί σε βρώμικη λέξη. Ε, λυπάμαι που οι πράσινοι υποστηρίζουν αυτές τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Οι τελευταίες εκλογές στην ε, Βουλγαρία ε, δεν κέρδισαν οι πράσινοι τίποτα στις εκλογές αυτές λόγω αυτής ακριβώς της τάσης γιατί οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος μόνο οι υπερασπιστές δεν είναι και οι ΜΚΟ πρέπει να πάνε φυλακή. Ενωτικής αριστεράς το λόγο έχει ο κύριος Κόκαλης για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Σε λίγες ώρες αυτή την αίθουσα θα κληθούμε να ψηφίσουμε να κηρύξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης. Ελπίζω να το κάνουμε, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει στον πλανήτη μας. Και το κάνουμε όχι για να προστατεύσουμε τον πλανήτη ή για να καταστρέψουμε τον πλανήτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το κάνουμε γιατί αυτή η έκτακτη ανάγκη αφορά την υγεία των ανθρώπων. Το κάνουμε για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και να αναγνωρίσουμε ότι το ανώτατο ανθρώπινο δικαίωμα είναι το δικαίωμα στην ανάσα και στο περιβάλλον εκείνο που μας επέτρεψε να εξελιχθούμε στα όντα που είμαστε σήμερα. τα τελευταίο, τελευταία χρόνια πάνω από πέντε άνθρωποι το χρόνο σκοτώνονται δολοφονούνται προστατεύοντας φυσικούς πόρους. αυτή η μάχη θα συνεχιστεί από κλιματικούς αγωνιστές κυρίως αυτόχθονες πληθυσμούς οι οποίοι προστατεύουν τη γη τους και προστατεύουν και εμάς τους ίδιους. Τα δάση τα προστατεύουμε γιατί μας προστατεύουν από την υπερέκθεση στο διοξείδιο του άνθρακα. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε δίπλα τους και στη Ρουμανία και στη χώρα μας και στο Λονδίνο και παντού θα βλέπουμε περισσότερους κλιματικούς αγωνιστές καθώς όλο και μειούμενοι πόροι υπάρχουν για όλο και περισσότερους ανθρώπους. Πρέπει να δημιουργήσουμε και εμείς μια γραμμή έκτακτης βοήθειας να παρέχουμε νομική υποστήριξη και να δημιουργήσουμε και ένα μηχανισμό άμεσης αντίδρασης στα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής εγγεγραμμένος είναι ο κύριος Σίντσης από τους μη εγγεγραμμένους, αλλά δεν τον βλέπω παρόντα στην αίθουσα. Επομένως, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μπεν Χούμπερ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο πρόσωπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ε, κατάσταση των υπερασπιστών του περιβάλλοντος ε, είναι όλο και πιο επίγουσα. Ε, βλέπουμε επίσης λίγα πράγματα στον τύπο, στην Αυστρία για παράδειγμα. Πολύ περισσότερες φωτογραφίες έχουμε από το πώς τη βάζονται ζώα στους τάβλους παρά πληροφορούμαστε για την τύχη πολλών υπερασπιστών του περιβάλλοντος και πρέπει να πω ότι οι αγρότες χρειάζονται δυνατότητες και βοήθεια για να αντιμετωπίσουν και την παράνομη υλοτομία και την αρπαγή γεών γιατί με την απερίμωση αφήνουμε να ε, δοθούν στη δημοσιότητα κάποια βίντεο τα οποία όμως παραπληροφορούν και αποπροσανατολίζουν. Πρέπει να δώσουμε τις ε, σωστές εικόνες. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε όχι τόσο τους υπερασπιστές ε, του περιβάλλοντος αλλά κυρίως τους υπερασπιστές των να υπερασπιστούμε τους αγρότες. Για 1,5 Ας ξεκινήσουμε, ξεκινήσουμε με τα καλά νέα. Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών συνειδητοποιεί ότι η σημασία των δασών είναι τεράστια και έχουμε διαχειριστεί με σχετικά αποτελεσματικό τρόπο τις δασικές εκτάσεις στην Ευρώπη και έχουν από τη δεκαετία του 90 τα δάση αυξηθεί σε μια επιφάνεια αντίστοιχη με το έδαφος της ελληνικής δημοκρατίας. Η δική μου χώρα, η Δανία, έχει επιλέξει να πολλαπλασιάσει τις δασικές εκτάσεις σε σχέση με το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά απαιτούνται και δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι καλό που έχουμε ένα νέο πρόγραμμα δράσης πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα προστατεύσει και τα πρωτογενή δάση αλλά και τη βιοπικιλότητα. Τμήμα του προγράμματος αυτού είναι να προστατεύσουμε φυσικά και αυτούς που προστατεύουν τα δάση και τη φύση. Δεν μπορώ, πως, δεν να πω σε αυτή τη φάση πώς αυτό μπορεί να γίνει, αλλά είναι σαφές ότι χωρίς αυτούς δεν θα πετύχουμε και απαιτείται να σεβαστούμε τους κανόνες με πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι μέχρι σήμερα. Απαιτούνται λοιπόν να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την προστασία και των δασών και αυτών που τα φροντίζουν. Ε, επόμενος ομιλητής εγγεγραμμένος είναι ο κύριος Γκερέρο, τον οποίον δεν βλέπω στην αίθουσα. Επομένως, το λόγο έχει η κυρία Βίσνιεύσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα δάση παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την καθαρότητα του αέρα που αναπνέουμε. Δεν χρειάζεται να σας πείσω γι' αυτό. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα βασικά γεγονός θα πρέπει να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις δασικές εκτάσεις. Υπάρχουν και καλά παραδείγματα και στην Πολωνία. Η Πολωνία όταν βλέπουμε την επιφάνεια των δασών ε, κάθε χώρα είναι στην κορυφή. 9 δις εκτάρια, το 30% της χώρας καλύπτεται από δασικές εκτάσεις. Τα περισσότερα από τα δάση αυτά ανήκουν στο κράτος και νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα διαχείρισης και αηφορίας. Κάθε χρόνο στην Πολωνία φυτεύουμε πάνω από 500.000 ε, φυτά, δένδρα. Και να υπογραμμίσω κάτι που είχε ε, ε, συζητηθεί και εδώ παλιότερα. Υπάρχει το δάσος της Βία που είχαν προκαλέσει ε, διαδηλώσεις, ε, η συζήτηση ε, για την κοπή των άρρωστων δένδρων. Και δυστυχώς αυτοί που προασπίστηκαν το περιβάλλον καταδίκασαν το δάσος. Χάσε 15 λεπτό το δάσος δεν έχει φωνή και οι γενναίοι άνθρωποι που το υποστηρίζουν και διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να το κάνουν. Θέλω να σας πω την ιστορία ενός Ρουμάνου ε, ακτιβιστή ε, του Γκάμπριλ Παό που είναι σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο διακινδύνευσε τη ζωή του προσπαθώντας να εμποδίσει να μετατραπούν τα δέντρα σε φθηνά έπιπλα. δέντρα τα οποία κόβονταν από το πάρκο των Δολομητών. Ε, ε, ε, το 2015 η μαφία των ξυλοκόπων ε, το έσπασε το κεφάλι, είχαν σκοπό να τον σκοτώσουν. Όλα είναι καταγεγραμμένα και πήρε στους εισαγγελείς τέσσερα χρόνια να στείλουν στα δικαστήρια τους ε, δράστες και πέρσι έκοψαν μεγάλα ε, δέντρα για να και, και έφτιαξαν τύχη για να τον εμποδίσουν να μαγνητοσκοπήσει την παράνομη δασοπονία την παράνομη συγγνώμη, υλοτομία. Τι θα κάνει η Κομισιόν για να προστατέψει τα δάση μας και το κόσμο που τα υπερασπίζει. Σπολτσάκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως η προστασία του περιβάλλοντος είναι σε ένα φυσικό πεδίο μάχης για την ανθρωπότητα. Θέλω να καταγγείλω τον, δολοφονία δύο υπερασπιστών των δασών στη Ρουμανία. Οι υπερασπιστές αυτοί ζουν και εργάζονται για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Πρόκειται για βιώσιμη ανάπτυξη ανάπτυξη και είναι και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, χειραγώγηση και κατάχρηση εξουσίας από πλευράς των δασοφυλάκων, ενώ δεν προβλέπεται καμία επιπλέον προστασία για τους ε, υπερασπιστές των δασών. Οι τοπικές κοινότητες υπερασπίζονται τους πόρους τους, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχουν κοινότητες στον κόσμο που αυτό το κάνουν με φυσικό τρόπο. Ε, και πραγματικά υπήρξε μια ε, αλλαγή στην δασοκομεία που έχει βελτιωθεί η κατάσταση δηλαδή στην Ευρώπη αλλά δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε στις, στις δάφνες μας. Ένα λεπτό. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια ε, παρατηρούμε αυξανόμενους αριθμούς διαμαρτυριών ε, προς υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιβαλλοντικοί ακτιβιστές όπως αυτοί στο δάσος ε, Μπιελοβιέσκα ή Count for Climate στην Πολωνία προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ανθρωπότητας και τα αιτήματά τους είναι καθηλωτικά. Όταν οι Πολωνοί διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για τις μαζικές, τη μαζική υλοτόμηση προστατευόμενων δασών ενημέρωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθήσει ο πύρη καθώς οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος παρενοχλούνται, συλλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αυτό που κάνουν. Εγώ ε, κάνω έκκληση να προστατευθούν τα δικαιώματα των, προστα... των υπερασπιστών των δασών και του περιβάλλοντος γιατί αυτοί είναι ροές και όχι εγκληματίες. Έχει ο κύριος Χόλμγκρεν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλο ένα και περισσότερες χώρες επιβάλλουν απαγόρευση για εγγραφή σε περιβαλλοντικές εργανώσεις. Αυτοί που αγωνίζονται υπέρ του περιβάλλοντος παρενοχλούνται, απειλούνται με ε, θάνατο και τρεις δολοφονίες την εβδομάδα σχετιζόμενες με το θέμα του περιβάλλοντος ε, ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να προστατευτούν τα δάση από την κλοπή ξυλίας ή από την παράνομη υλοτόμηση. Η φύση πρέπει να προστατευθεί. θα πρέπει να προστατευτούν και οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριο Μορέλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίως η αποκατάσταση και η προστασία των ευρωπαϊκών δασών είναι μεγάλη πολιτική ε, πρόκληση. Όμως ε, θα πρέπει να πάψουμε να είμαστε υποκριτές γιατί ναι, προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά δάση αλλά εξάγουμε την ε, αποψήλωση των δασών, την, υπογράφοντα συμφωνίες συνεργασίας όπου δεν προβλέπεται τίποτα και μάλιστα πρόκειται για πρωτογενή δάση, ας πούμε η συμφωνία με το Βιετνάμ ή η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί με το Μερκοσούρ που είναι στην ουσία μια παρότρινση για την αποψήλωση των δασών. Υπάρχουν και κοινωνικά διακυβεύματα, γιατί μιλήσαμε για τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος που αυτή τη στιγμή θεωρούνται εγκληματίες και πολλές φορές διώκονται, αλλά και για τους εργαζόμενους στο δάση, για την, ε, για την δασοκομεία, την... Ε, ε, καλλιέργεια των δασών που ζουν με ιδιωτικοποίηση. Ας πούμε στη Γαλλία το, η Εθνική Υπηρεσία των ε, Δασών, αυτοί οι εργαζόμενοι, οι δασονόμοι, οι δασοκόμοι πρέπει να προστατευτούν. Και επίσης πιστεύω θα πρέπει να έχουμε πιο καλό συντονισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών. Έχουμε ένα σωρό κείμενα. Θα έπρεπε να φτιάξουμε λοιπόν ένα νομοθετικό πακέτο για τα δάση, ομοιόμορφο, ε, που θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία της γεωργικής πολιτικής και της ανάπτυξη των βιοκαλλιεργειών αυτό λοιπόν είναι ένα εργοτάξιο το οποίο θα πρέπει να μπει μπροστά γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω γεννηθεί περιτριγυρισμένος από καστανιές βελανιδιές ε, στην ε, χώρα μου, όπως και παντού τα δάση είναι πνεύμονες ζωής και ήταν ε, πηγή θαλπορής, τροφίμων για αιώνες τα δάση και προστασίας. Πρέπει σίγουρα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας ε, στους δασοφυλάκες στη Ρουμανία που ε, πλήττονται όπως επίσης ε, και σε όλους όσοι προσπαθούν να απερασπιστούν το περιβάλλον. Θα πρέπει τα αυτόχθονα πρωτόγωνα δάση να τα υπερασπιστούμε γιατί από την λεμαργία και την απληστία κινδυνεύουν αυτά τα δάση ε, υπάρχουν αυτές οι δασικές μονοκαλλιέργειες ε, που ουσιαστικά φτωχαίνουν το έδαφος ε, και διευκολύνουν και το έργο των εμπριστών στη θέση των ε, δασών. Θέλουμε να στηρίξουμε και την αναδάσωση αλλά και την ε, εργασία αυτών οι οποίοι ε, είναι υπεύθυνοι για την δασοκομεία. Διότι ένα δάσος αρχαίγωνο ουσιαστικά είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Το επενθυμίζω αυτό. Ευχαριστώ. υπάρχει κύριε Γκονσάλες, μία μπλε κάρτα από τον κύριο Μπούντα. Τη δέχεστε. You have a blue card from Mr. Buddha. Do you accept it? Mr. Buddha. 30 seconds for a question. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l întreb pe distinsul coleg dacă este de acord cu ceea ce... Έχω μία ερώτηση για τον αγαπητό συνάδελφο. Δεν θα ήταν καλό από εδώ και πέρα τα δάση στη Ρωμανία και οι υπερασπιστές τους να έχουν όπλα για να μπορούν να προστατεύουν τους εαυτούς τους. Ε, μήπως θα πρέπει να γίνει αυτό για όλους τους εργαζομένους. Νομίζω ότι η κατάσταση στη Ρωμανία είναι ιδιαίτερα είναι διαφορετική από ό,τι αλλού. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια λύση για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν ε, φυσικά να είναι εξοπλισμένα με συστήματα προστασίας νόμιμα. Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών προχωρούμε στη διαδικασία του Catch Έχω δεχθεί έξι αιτήματα, τα κάνω και τα έξι αποδεκτά. Το λόγο έχει η κυρία Σόντροβα για ένα λεπτό. You have the Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο γιατί θέλω να αναφέρω δύο-τρία πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, στην επόμενη θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη επισταμένως ε, να προβούν σε αναδασώσεις. Διότι ναι μεν υπάρχουν ακόμη αρκετά μεγάλες δασικές εκτάσεις, αλλά έχει υποβαθμιστεί ποιότητά του λόγω των περιόδων ξηρασίας, της κλιματικής αλλαγής ε, και άλλων προβλημάτων, ζυζανίων κτλ. Θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν ε, τους δασοκόμους και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες αναδάσωσης. Επίσης, στην Τσεχία υπάρχουν εκατοντάδες ε, άνθρωποι που προσπάθησαν να αναδασώσουν χιλιάδες εκτάρια και αυτούς πρέπει να τους επενέσουμε γιατί αυτό δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον και γι' αυτό και δεν θέλω να συμφωνήσω ε, και με την προσέγγιση του πρώτου της Βραζιλίας και τον τρόπο που αντιμετώπισε το πρόβλημα ε, στη χώρα του. ο κυρίος Τούσκ ήθελε να παρασχεθεί βοήθεια στον Πολσονάρο, αλλά δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό αν δεν τηρούν τα σχετικά. κύριος Mr. you have the floor. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που αναφέρθηκαν στη χώρα μου, στη Ρωμανία. Κλέγουν τα δάση στην ε, ε, Ρωμανία γιατί κάθε ώρα και στιγμή εκτάρια δασών εξαφανίζονται. Στη Ρουμανία, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθεί να μειώσει τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακος. Δυστυχώς η προστασία είναι ανεπαρκής και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που αναφέρθηκε στα της Ρουμανίας. Μερικές φορές οι εθνικές πολιτικές ε, στις χώρες μας δεν προστατεύουν με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Νομίζω ότι για όλες αυτές τις απώλειες δασικών εκτάσεων σήμερα θα χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια για την αναπλήρωσή τους. Η γενιά μας θα πρέπει να συντηρήσει σε καλή κατάσταση τα δάση. Ας δώσουμε λοιπόν στα δάση τη σημασία που τους αξίζει. Το λόγο έχει η κυρία Κονέτσινα για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλές φορές ασκούμε κριτική ε, σε χώρες εκτός Ένωσης ε, για την αποψήλωση των δασών. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ, ε, στην Ένωση, το πρόβλημα. Δυστυχώς γιατί και εδώ βλέπουμε να ε, διακυβεύονται ζωές. Έχουμε την μαφία του ξύλου που ε, οδήγησε ε, στην απώλεια της ζωής δύο Ρουμάνων δασοφυλάκων. Αυτό πραγματικά για μένα είναι αποτροπιαστικό. Να γίνεται εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πατρίδα μας. Επίσης, το ότι κάθε μέρα 9 εκτάρια αρχαίων δάσου στη Ρουμανία αφανίζονται. Εμείς καθόμαστε δε με σταυρωμένα χέρια. Είναι κάτι που επίσης ε, με σοκάρει. Η Συμφωνία των Παρισίων δεν είναι ένα χαρτί ε, και στην πράξη δεν σημαίνει τίποτα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να την επιβάλλουμε, αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε μπορούμε να κηρύσουμε σε όλους τους άλλους πρέπει να κάνουν και εμείς να μην μπορούμε να βάλουμε τον οίκο μας σε τάξη πρέπει να καταδικάσουμε αυτά που έγιναν στη Ρουμανία, κύριε Πρόεδρε, και σα ε, παρακαλώ να λάβετε συγκεκριμένα μέτρα για να αποτραπούν όχι μόνο βέβαια οι δολοφονίε, αλλά η απώλεια ενό πολύτιμου φυσικού πόρου που είναι τα δάση μα. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπτήρε στι οικογένειε των ε, δύο δασοφυλάκων. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Θέλω να καλέσω όλους τους ευρωβουλευτές, κυρίως τους 20 που είμαστε εδώ παρόντες, να φροντίσουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Ο συνάδελφος μίλησε για τη μαφία της ε, υλοτομίας και υπάρχει και στην Κροατία. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Τρεις δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία μας, έχουμε 500 ε, ε, εκτάρια τετραγωνικά εκτέρια. Δηλαδή, όμως ε, η υλοτομία προχωρά πολύ γρήγορα και η παράνομη υλοτομία επίσης. Δηλαδή, πέρα από την νόμιμη έχουμε και την παράνομη. Και αυτά γίνονται τώρα, είναι εκτιμήσεις. Δεν υπάρχει σχεδιασμός ε, όσον αφορά την υλοτομία ε, και η ξυλία αυτή στέλνεται παράνομα και σε άλλες χώρες. Η κροατική βιομηχανία ποτέ δεν είχε τέτοιες δυσκολίες. Ε, να βρει ξύλο, ε, να βρει ξυλία. Η Κροατία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτό το πρόβλημα και να τα βάλει με τη μαφία. Γι' αυτό ε, πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τα δάση. You have the floor for one minute. Λίγα λόγια στα φιλανδικά. Θα πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλές χώρες όπου η προστασία των δασών, η βιοπικιλότητα είναι πολύ σημαντικό και η βιομηχανική, η οικονομική χρήση των δασών είναι βιώσιμη. Η Φιλανδία είναι ένα παράδειγμα υποδειγματικό. Προστατεύουμε με ένα σωρό στάνταρ τα δάση μας. 400.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους. Λίγο παραπάνω από την όλη έκταση της Δανίας έχουμε. Έχουμε καταφέρει όμως να τα συντηρούμε και να κάνουμε βιώσιμη εκμετάλλευση των δασών μας. Μπορούν αυτά τα δυο να συμβαδίσουν. Μπορούν να γίνουν πολλά για την προστασία των δασών, για να γίνει βιώσιμη χρήση των δασών. Αυτά τα δυο θα πρέπει να συμβαδίσουν. Και κύριος για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόσφατη δολοφονία δύο Ρουμάνων δασοφυλάκων τονίζει την ανάγκη να προστατευθούν οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος στην Ευρώπη και να σωθούν τα τελευταία φυσικά δάση της Ευρώπης. Το 2018 δολοφονήθηκαν ακτιβιστές και εκατοντάδες ακόμα φυλακίστηκαν στην Ινδία, στη Βραζιλία, στην Κολομβία, στην Ινδονησία. Πρέπει να ε, περιληφθεί υποχρεωτικά στα ανθρώπινα δικαιώματα για τις εταιρείες και τα, και ε, χρηματοπιστωτικά όργανα που παρέχουν τέτοιες ε, υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι υπόλογες για τις δραστηριότητε των ε, παραρτημάτων τους στις χώρες εκτός Ένωσης. Υπάρχει μεγάλη κατάχρηση και αποψήλωση των δασών στη Βραζιλία αυτή τη στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνένοχη λόγω των εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει με τη Βραζιλία και που αυξάνει, ε, αυξάνουν την υλοτόμηση. Όχι μόνο θα εξαφανιστούν οι μικρές ε, ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη, αλλά θα καταστραφούν και τα δάση στην Βραζιλία. Το λόγο, το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής ο Επιτροπός κ. Μίμητσα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Η σημερινή συζήτηση ήταν πολύ σημαντική. Συμφωνούμε όλοι. Πρέπει να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε τα δάση στον πλανήτη. Πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τους κλιματικούς αγωνιστές που τόσο θαραλέα ύψωσαν το ανάστημά τους για να προστατεύσουν τη φύση πράγματι. Οι κλιματικοί αγωνιστές είναι απαραίτητη σύμμαχή μας στην προσπάθεια της πρόθεσης των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Θέλω να ποτέ σοφόρο τιμή ε, στους ε, προσφάτους δολοφονηθέντες ε, Πόπ και Κορτσογκοάγια, τους δύο Ρουμάνους δασοφύλακες και να εκφράσω τα θερμά ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Σίγουρα θα αξιολογήσουμε την ανάγκη λήψης νέων ρυθμιστικών μέτρων, αλλά Ήδη θα πρέπει ε, αποτελεσματικά να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε. Ε, επιβάλλει. Και σίγουρα οι αρχές, οι εθνικές έχουν ευθύνη. Πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουμε την ε, πραγματική εφαρμογή και της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας επιτόπου. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές περιλαμβανομένης και της Ρουμανίας ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή και επιβολή της νοσιακή νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση έληξε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού ε, και το θέμα είναι η κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο πρώτος εκ των συντακτών, ο κύριος Ραφαέλ Γκλουξμάν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, από τότε που έγινα βουλευτής... Ασχοληθήκαμε με πάρα πολλές χώρες αλλά δεν ασχοληθήκαμε καθόλου για την επανάσταση η οποία έγινε την επόμενη, στην απέναντι όχθη στην Αλγερία. Εκατομμύρια Αλγερινοί άνδρες και γυναίκες εδώ και εννέα μήνες διαδηλώνουν με δημοκρατία δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς ε, για την καταστολή και τη βία δεν έχουμε πει κουβέντα και τα βασανιστήρια επίσης Πρόκειται για μια συνένοχη σιωπή. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει. Πρέπει να περάσει το ψήφισμα αυτό αλληλεγγύης. Είναι το τέλος μιας τεράστιας αδικίας. Πρέπει να δείξουμε ότι στηρίζουμε τον λαό της Αλγερίας. Όπως λένε στην οικογένειά μου, one, two, three, viva l'Algérie. Συντάκτες είναι ο κύριος Μπέργκ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατεκπρόσωπε, τους τελευταίους μήνες η αλγερινή κυβέρνηση έχει κλείσει με βίαιο τρόπο οκτώ προστατικές εκκλησίες τουλάχιστον. Υπάρχουν μικρές χριστιανικές κοινότητες στην Αλγερία που διώκονται και υπάρχει η ε, βλασφημία ε, που θεωρείται δηλαδή αδίκημα να μπορεί κανείς ε, να ασκεί τη λατρεία του, τη χριστιανική. Πολλοί φυλακίζονται που δεν, κάνουν, ε, δεν ακολουθούν το Ραμαζάν για παράδειγμα. Έχουμε τέτοια στοιχεία που μπορούν να δείξουν ότι πραγματικά υπάρχει δίωξη των χριστιανών το 20% ήταν χριστιανοί ε, στην ε, Μέση Εγγύη Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική πριν από 20 χρόνια και τώρα είναι μόνο 4%, μάλλον πριν 100 χρόνια και τώρα είναι μόνο 4%. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η προσπάθεια να διερευνηθούν οι λόγοι και οι συνθήκε υπό τι οποίε διώκονται οι χριστιανοί. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει μια τέτοια πρωτοβουλία. Θα πρέπει να μπορούν οι χριστιανοί χριστιανοί χωρίς φόβο, ε, χωρίς ε, να φοβούνται ότι θα υποστούν διάκριση, απειλές, τα λοιπά, να μπορούν να ασκούν ε, την λατρεία τους και να καταρριχθεί σχετική νομοθεσία. Βαντάλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια στην Αλγερία είδαμε πραγματικά το άσχημο πρόσωπο του καθεστώτος. Ένα πρόσωπο καταστολής ένα πρόσωπο έλλειψης ε, ανοχής, καταστράφηκαν εκκλησίες, έκλεισαν εκκλησίες. Στις 16 Οκτωβρίου στο ουζού έγινε μια επίθεση σε εκκλησίες και τραυματίστηκαν πιστοί. Και από τον Ιούνιο του 16 μέχρι τον Ιούνιο του 18 Ε, διώχθηκαν και πολλοί αλμάντι όπως λέγονται χριστιανοί στην ε, ε, Αλγερία. Η έκθεση της υπηρεσίας της διπλωματικής λέγει ότι η κατάσταση στην Αλγερία παραμένει κρίσιμη και είναι μια κατάσταση προσπάθειας περιορισμού της θρησκευτικής ελευθερίας θα πρέπει οι πιστοί να μπορούν να συγκεντρώνονται σε εκκλησίες και σε άλλους τόπους λατρείας. Δυστυχώς όμως στην Αλγερία όπως και σε άλλες χώρες της περιοχής τα δικαιώματά τους ε, παραβιάζονται συστηματικά. Είχα δύο λεπτά. Ε, συνεπώς λοιπόν θα πρέπει η κυρία Μογκερίνη να διαμαρτυρηθεί για την απαράδεκτη κατάσταση στην Αλγερία και οι εκκλησίες οι οποίες έκλεισαν πρέπει να ξανανοίξουν. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να εμπλακεί και η ειδική εκπρόσωπος για τα θέματα των ελευθεριών. Επίσης συντάκτης. Monsieur le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 Λοιπόν. Γκετά λέγομαι κύριε Πρόεδρε. Ας φανταστούμε, ας φανταστούμε ότι αυτό το τεράστιο κίνημα που αναταράζει την Αλγερία σήμερα, νέοι οι οποίοι προσβλέπουν στην αξιοπρέπειά τους, το κράτος δικαίου και την αξιοπρέπεια, ας φανταστούμε μόνο πως αυτό το κίνημα ε, και θα νικήσει. Δεν θα ήταν μόνο θέμα περηφάνειας Αλγερίας, θα ήταν ε, η δικαίωση της κινητοποίησης όλης αυτής της ενέργειας υπέρ των δικαιωμάτων του Μαγκρέπ, της συνεργασίας, της οικονομικής και της πολιτικής πολιτιστικής με την Ευρώπη και το τέλος της ε, ε, υστέρησης ε, των χωρών του Μαγκρεμπ. Θα ήταν προς όφελος όλων μας, Μαγκρεμπίνων και Ευρωπαίων και γι' αυτό πρέπει να υιοθετήσουμε αυτό το ψήφισμα κατά μια αβάσαχτης και παράλογης καταπίεσης που μπορεί να διαλύσει αυτό το αλγερινό όνειρο. Ας δώσουμε την ελπίδα και την στοργή της Ευρώπης στους Αλγερινούς. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Βέιμερς για ένα λεπτό. Tack, ε, herr talman. Tidigare i höst ε, röstades förslaget om att debattera kyrkostängningarna ner utav... Υπήρξε μια συζήτηση λίγους μήνες πριν σχετικά με το κλείσιμο τόπων λατρείας στην Αλγερία και η συζήτηση αυτή συγγνώμη έγινε στο Κοινοβούλιο της Σουηδίας και χαίρομαι που επανέρχεται η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό, δεν μπορούμε παρά να εμείνουμε στην ελευθερία άσκησης ε, της θρησκευτική πίστης. Και λυπάμαι που αφαιρέθηκε ο τίτλος, ε, το τμήμα ε, για τη θρησκεία και δεν είναι πρώτη φορά, η αριστερά ε, προσπαθεί συστηματικά να αποκρύψει τις θρησκευτικέ διώξεις. Θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουμε τις διώξεις εις βάρος των χριστιανών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έστειλε ένα εκατομμύριο κουρώνες, λέει ομιλήτρια, στην Αλγερία μέσα σε πολύ λίγα χρόνια και ταυτόχρονα οι αρχές της Αλγερίας συνέχισαν και εντατικοποίησαν τις διώξεις εις βάρος των χριστιανών. Οι εκκλησίες κλείνουν και οι σύλλογοι των χριστιανών δεν αναγνωρίζονται. Αυτό είναι αντίθετο με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι αντίθετο και με το ίδιο το συνταγματικό χάρτη της Αλγερίας και πρέπει να πιέσουμε τη χώρα αυτή να σταματήσει των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λόγο έχει ο κύριος Μάντλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Πριν από μια εβδομάδα είχα την ε, ευκαιρία στη δική μου ε, πατρίδα, στη Βιέννη, να μιλήσω ε, για τις ε, μουσουλμάνους ε, που είχαν οργανώσει μια σχετική συνάντηση και για την θρησκευτική ελευθερία εκεί. Τώρα μιλάμε εδώ για την ελευθερία εκφρασής. Έχουμε ένα happy hour εδώ και μιλάμε όλοι. Ο Ντάμιαν με την Ειρήνα από το και ο κύριος Μπελαμή από, την, από το ΕΛΚΑ και άλλοι. Γιατί το το λέω αυτό γιατί Αυτές τις οικουμενικές αξίες ε, τις έχουμε εμείς εδώ ε, θεμελιώσει. Θέλουμε την ελευθερία ε, έκφρασης, τη θρησκευτική ελευθερία να την υπερασπίσουμε και να αναφέρουμε έτσι με δυνατή φωνή πράγματα που συμβαίνουν. Παραδείγματο χάρη στην Αλγερία για αυτή την μειονότητα των μουσουλμάνων οι οποίοι μόνο και μόνο γιατί θέλουν να τη λατρεία τους τιμωρούν Υπάρχουν εκκλησίες ε, που κλείνουν, ε, όπως και οργανώσεις ε, γυναικείες. Έχουμε εκλογέ στις 12 Δεκεμβρίου στην Αλγερία. Θα πρέπει οι Αλγερινοί να πάρουν τις σωστές αποφάσεις εκείνη τη μέρα. ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχει η κυρία Αρένα για ένα λεπτό. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και πάνω από εννέα μήνες οι Αλγερινοί ε, συγκεντρώνει το θαυμασμό του κόσμου λόγω ε, των δημοκρατικών τους ε, επιδιώξεων που εκδηλώνονται με ειρηνικό τρόπο αλλά με αποφασιστικό τρόπο. Η Αλγερία έχει υπογράψει διάφορες διεθνείς συνθήκες μεταξύ αυτών και την Παγκόσμια Δήλωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το σύμφωνο που σχετίζεται με τα πολιτικά και δικαιώματα για να σας αναφέρω έτσι κάποιες συμβάσεις. Έπειτα υπάρχουν και εγγυήσεις στο Σύνταγμα της Αλγερίας. Ωστόσο, προσωπικότητες βρίσκονται αυτή τη στιγμή υποκράτηση επειδή εξέφρασαν ε, μία επιθυμία υπό την ε, ε, δικαιολογία ότι αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Μέσα από το ψηφίσμα μας εμείς καλούμε τις αρχές της Αλγερίας να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και τους κρατούμενους συνείδησης. Πρέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία έχει υπογράψει η Αλγερία να είναι εγγυημένα, ιδιαίτερα η ελευθερία λόγου και η ελευθερία του συνέχεια έρχεστε. Ε, η Ευρώπη είναι φίλη όλων των Αλγερινών, ανδρών και γυναικών και ε, πρέπει να τιμήσουμε την εταιρική σχέση την οποία υιοθετήσαμε τον Μάρτιο του 2017 και όπου ε, αναλάβαμε την υποχρέωσή μας να σεβαστούμε τις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Renew Europe, το λόγο έχει για ένα λεπτό επίσης ο κύριος Μπένιον. Uh, thank you, Chair. Uh, the democratic process... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δημοκρατικέ διαμαρτυρίε στην Αλγερία φαίνεται να έχουν επιτύχει το στόχο του. Όταν ο πρόεδρο Μπουτεφλίκα αντέστρεψε την απόφασή του να είναι υποψήφιο για πέμπτη διαδοχική θητεία τον Απρίλιο φέτο. Ωστόσο, οι ηγέτε των διαφόρων κινημάτων διαμαρτυρία έχουν ε, ωστόσο παρατηρήσει ότι πρόκειται για ένα καθεστώς το οποίο αντικαθιστά τον Μπουτεφλίκα που και φαίνεται να είναι στρατιωτικό ε, το καλύτερο θα ήταν η Αλγερία να, προσε... να προσεγγίσει το Μαρόκο και την Ισία και να ανοιχτεί περισσότερο στον κόσμο. Εκφράζω ε, δε και εγώ τις ανησυχίες όπως και οι συνάδελφοι για τις ε, θρησκευτικές ελευθερίες και όταν πια θα γίνουν αυτές οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν ελεύθερα και δίκαια. Και έπειτα θα ήθελα να δω την Αλγερία να ανοίγει τα σύνορά της προς Μαρόκο και προς την Ισία, ώστε να υπάρξει μια ένωση Μαγκρέμπ που θα λειτουργήσει ως ένας ισχυρό εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε με οικονομική ανάπτυξη που θα φέρει ε, ευημερία και ειρήνη στην περιοχή του Μαγκρέμπ. Πρασίνων, το λόγο έχει η κυρία Γεμπού για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ομάδα των Πρασίνων αποφάσισε να στηρίξει, ε, να καταθέσει ένα ψήφισμα στα επίγοντα για τους εξής λόγους. Επιλογή πολιτική πριν από τις εκλογές της 10 ε, Δεκεμβρίου. Ο κίνδυνος να πολιτικοποιηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να υποβαθμιστεί η αξιοπιστία της αντιπολίτευσης και των Αλγερνών που διαδηλώνουν εδώ και 9 χρόνια. Ο κίνδυνος να τροφοδοτηθεί η προπαγάνδα των αρχών για εξωτερική παρέμβαση. Ε, είναι σημαντικό να στηριχθούν οι Αλγερινοί ε, με σταθερό τρόπο Παρά, τις, παρά τις διάφορες ε, επιφυλάξεις, είμαστε υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Η στήριξή μας στον Αλγερινό λαό δεν θα σταματήσει εδώ. Ε, είμαστε κινητοποιημένοι στο πλευρό του αλγερινού λαού για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του και χαιρετίζουμε την υποδειγματική συμπεριφορά του αλγερινού λαού ε, που, ήταν, που είναι εξαιρετικά ειρηνική και έπειτα θέλουμε ε, τέλος ο αλγερινός λαός να αποφασίσει μόνος του. Και όπως λέμε στο σπίτι μου και στην Αλγερία ταχεία Ζαζάιρ. δηλαδή ζήτω η Αλγερία. ότι βρισκόμαστε στον κύκλο των ημιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, στη διάρκεια του οποίου δεν προβλέπονται μπλε κάρτες και γι' αυτό δεν έχει ενεργοποιηθεί και στην ηλεκτρονική διαδικασία η δυνατότητα υποβολής τέτοιου αιτήματος. Επομένως, όταν ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο, θα ενεργοποιηθεί αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τον κανονισμό. Προχωρούμε στην ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ο κύριος Κολάρ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ne peut laisser personne αυτό που συμβαίνει στην Αλγερία δεν μπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο για δύο λόγους. Ο πρώτος βασίζεται σε αρχές και ο δεύτερος βασίζεται στην πραγματικότητα. Οι αρχές λέγουν ότι οπουδήποτε παραβιάζονται οι ελευθερίες θα πρέπει να δράσουμε για να τις υπερασπιστούμε. Η πραγματικότητα είναι δάκρυα, πνιγυρή ατμόσφαιρα, αίμα πολλές φορές και απελπισία και το γεγονός ότι ανάμεσα στη Γαλλία και την Αλγερία υπάρχουν σύνδεσμοι πολιτικοί, οικονομική, κοινωνικοί, συναισθηματικοί και όταν ο κόσμος δεν πάει καλά στην Αλγερία την εγκαταλείπουν οι κάτοικοί της και έρχονται στη Γαλλία η οποία όχι δεν θέλει αλλά δεν μπορεί εν να τους φιλοξενήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εγκρίνουμε το συγκεκριμένο ψήφισμα εξ ονόματος των ελευθεριών, εξ ονόματος των αρχών και, ονόματος της, και εξ ονόματος της ίδιας μας της ύπαρξης. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ρούισεν. Dank u wel, voorzitter. Geachte collega's, de berichten die ons bereiken uit Algerije waren ons grote zorg. Η έκθεση αυτή για την Αλγερία περιλαμβάνει στοιχεία που μας ανησυχούν όλους και δεν αναφέρομαι μόνο στις διαδηλώσεις. Ανησυχώ και ανησυχώ επίσης και για την ελευθερία της θρησκευτική λατρείας. Επαναλαμβάνω ότι έχουν κλείσει οι εκκλησίες και οι πιστοί έχουν με βία απομακρυνθεί από τον τόπο λατρεία τους. Η τέταρτη παράγραφος περιλαμβάνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις αρχές της Αλγερίας, λέγοντας ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Η εταιρική μας σχέση με την Αλγερία, στα πλαίσια επίσης και της Euromed, θα μας δώσει την ευκαιρία να επανέλθουμε με έντονο τρόπο στα θέματα της ελευθερίας άσκησης της θρησκευτική πίστης. Νομίζω ότι η κυρία Μογκερίνη θα χρησιμοποιήσει τις επαφές της με τις αρχές της Αλγερίας έτσι ώστε να εξηγήσει σωστά την κατάσταση. Σόιντροβα, ένα λεπτό. Χθε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν μια μέρα που είναι αναγνωρισμένη διεθνώ αφορά τη δίωξη των χριστιανών λόγω της ε, θρησκείας τους. Η Αλγερία είναι στην 122η θέση από τις χώρες που διώκουν τους χριστιανούς. Και το Υπουργείο έκλεισε πέντε προστατικές εκκλησίες και έχοντας τις παράνομες εκκλησίες γίνονται αντικείμενο επιθέσεων στη διάρκεια της λειτουργίας εμείς ζητούμε το Υπουργείο Εσωτερικό να εγκρίνει την ε, ίδρυση και τη λειτουργία ε, των ε, χριστιανικών οργανώσεων ε, να φυλάξει την θρησκευτική ελευθερία, γιατί αυτό κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι γιατί βλέπω ότι υπάρχει ε, υπερκομματική υποστήριξη σε αυτή την υπόθεση. Το λόγο έχει η κυρία Ρίση, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωτεκπρόσωπο. Το αλγενό Καθεστώ καταστέλει συγγνώμη, της ελευθερίας. Από τις 22 Φεβρουαρίου το λαϊκό ε, κίνημα ε, Χαρίκ έχει πλέον καλύψει όλη την ε, χώρα, κατεβαίνουν όλοι στους δρόμους. Έχουμε τις προεδρικές εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου, κάτι το οποίο όρισε μάλιστα ο στρατός. Καταπιέζει τα δικαιώματα των ε, συνδικαλιστών, των δημοσιογράφων, των φοιτητών, των εργατών. Εδώ και 10 μήνες έχουν κατέβει όλοι αυτοί στους ε, δρόμους. Υπάρχουν 42 διαδηλωτές που καταδικάστηκαν σε εξάμεινη κάθερξη επειδή ε, σήκωσαν ένα ε, λάβαρο των βερβέρων και βλέπουμε ότι μόνο και μόνο γι' αυτό ε, καταδικάζονται. Αυτό δείχνει ότι έχει ολιστήσει σε αυταρχισμό το καθεστώς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν. τα Ναι, ζητούμε την ελευθερία για τον αλγερινό λαό. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ντρεώστο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε. Με λυπεί που διαπιστώνω ότι αποσύρθηκε από το τίτλο από τον τίτλο αυτού του ψηφίσματος η ανεξιθρησκεία. Λες και η θρησκεία είναι ταμπού. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε ανοιχτά να μιλήσουμε για θρησκευτικέ διώξει και κυρίω για αυτέ εναντίον των χριστιανών. Θυμίζω πω η Αλγερία είναι η 22η χώρα στον κόσμο που είναι πιο δύσκολο να είναι κανείς ε, χριστιανός. Να θυμίσουμε μόνο ότι τον Οκτώβριο ότι η αλγερινή ειναι κανει χριστιανο να θυμισουμε μονο οτι έκλεισε τρει εκκλησίε και την πιο μεγάλη τη χώρα. Και συχνά τα θύματα των διώξεων είναι χριστιανοί χριστιανοί που έχουν ε, αξιοπιστήσει από το Ισλάμ. Ε, για μας η ανεξιθρησκεία είναι ένα θεμελιώδες ε, δικαίωμα, των ανθρώπινο δικαίωμα. Δυστυχώς διώκονται οι χριστιανοί και θα αναφέρω τα λόγια του, του Πάπα Βενέδικτου 16 όταν λέει ότι ε, η σημασία η κοινωνική της θρησκείας είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μην αφαιρεθεί αυτή η, λόγια, αυτή η λέξη ανεξιθρησκεία και να κρυφτούμε πάλι πίσω από μια πολιτικό ορθή ορολογία. Που έχει ο κύριος Μπουξαντέ για ένα λεπτό. Μας ανησυχούν τα νέα τα οποία έρχονται από την Αλγερία, οι καταστολές των διαδηλώσεων, η δίωξη συγγραφέων, η δίωξη ε, δημοσιογράφων και ο περιορισμός της θρησκευτική ελευθερίας και η διώξηση εις βάρος των χριστιανών. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να παίρνουμε αποτελεσματικές αποφάσεις ε, και να μην προκαλούμε καταστάσεις και αλλαγές όπως αυτές που επισυνέβησαν στη Λιβύη και στη Συρία και που οδήγησαν τις χώρες αυτές σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι στο παρελθόν. Το θέμα δεν είναι να λύσουμε μόνο τα θέματα της Αλγερίας, αλλά η Αλγερία θυμίζω ότι είναι μία από τις χώρες η οποία συνεισφέρει ε, περισσότερο θα έλεγα από άλλες στην αποστολή σε εισαγωγικά παράνομων, ε, παράτυπων μάλλον μεταναστών που φεύγουν από την Αλγερία και φτάνουν κυρίως στην περιοχή της Αλμέρια στην Ισπανία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της μεταναστευτικής πολιτικής. Ο κύριος Ριβιέρα. από το 1830 μέχρι το 1962 ήταν μια χώρα η Αλγερία με θρησκευτική ελευθερία χριστιανοί, εβραίοι και μουσουλμάνοι μπορούσαν να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα χωρίς καμία ανάγνωση ε, φανατική. Αλλά από το 62 με την ηγεσία του Εφελέν διώκονται οι μειονότητες οι εβραϊκές και οι χριστιανικές και οδηγούνται στην εξαφάνιση. Το να έχει κανείς τη βίβλο στην τσάντα του σημαίνει πέντε χρόνια φυλάκιση οι διάφορες κυβερνήσεις ε, επιτρέπουν να βανδαλίζονται φυσικά τα νεκροταφεία, τα εβραϊκά και τα χριστιανικά. Η Αλγερία εδώ και 30 τουλάχιστον χρόνια ε, κυμαίνεται ανάμεσα στον, στην τρομοκρατία την τζιχαντιστική και σε μια κατασταλτική αυστηρά κυβέρνηση. Νομίζω ότι μόνο με την αλλαγή της διεφθαρμένης εξουσίας θα μπορέσουν να αλλάξουμε. Ομιλητών, προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί 7 αιτήματα. Επειδή τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά με το χρόνο, θα κάνω και τα 7 αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριος Πόλτσακ για ένα λεπτό. pane předsedo. <clears throat> já bych chtěl samozřejmě rovněž odsoudit násilí ke kterému dochází. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θέλω να καταδικάσω τη βία που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες στην Αλγερία. Βλέπουμε τεράστιες διαδηλώσεις στη χώρα. Καθώς η κυβέρνηση καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχουμε δώσει τη δεύτερη προσοχή στην αλλεργία κατά το παρελθόν. Θα πρέπει ξεκάθαρα να καταδικάσουμε την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα βασανιστήρια, τη βία Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Υπάρχει βία και σε βάρος των μειονοτήτων και ιδίω των χριστιανικών. Εξ όσων γνωρίζω, εμείς υποστηρίζουμε με, την, ε, με αναπτυξιακή βοήθεια την Αλγερία τις προηγούμενες δεκαετίες. Πολλά έχουμε δώσει, πολλά χρήματα στη χώρα, άρα περιμένουμε να πληρούνται κάποιοι κανόνες, ε, υπάρχουν όροι που θα πρέπει να τηρεί η χώρα. Καλό λοιπόν την είπατε εκπρόσωπο να φροντίσει ε, η αναπτυξιακή αυτή βοήθεια να δίνεται υπό όρους και προϋποθέσεις. Ευχαριστώ. Λόπεθα Γιλάρη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά ε, και είναι σημαντικό να συζητούμε την Αλγερία και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Διπλωματία για να προωθήσει τη δημοκρατία και τα δικαιώματα εκεί όπου υπάρχει καταστολή βία παρατεταμένη. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όταν άρχισε να εφαρμόζεται το δίκαιο εκεί ε, στην Αλγερία μέχρι το 1962 ε, η Αλγερία κέρδισε την ανεξαρτησία της μετά, αλλά ε, ε, ξέρουμε ότι υπήρξε αυτό το στρατιωτικό καθεστώς για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε αυθαίρετες κρατήσεις και μαζικές συλλήψεις αντιφρονούντων ουσιαστικά για να μην γίνουν εκλογές. Οπότε φλήκα μετά από 30 χρόνια επιτέλους κάποια στιγμή ε, κατάλαβε ότι δεν πρέπει να ξαναυποβάλει υποψηφιότητα και ήταν αρχικά η ημερομηνία των εκλογών 4 Ιουλίου μετά πήγε ε, το Σεπτέμβριο και τώρα 12 Δεκεμβρίου. Δεν έχουν γίνει ακόμη γιατί η προσπάθεια είναι να κατασταλεί η αντιπολίτευση και οι αντιφρονούντες να μην μπορέσουν να ε, διεκδικήσουν τίποτα. Πρέπει να προωθήσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα για και την δημοκρατία, για να είναι επιτέλους αυτά πραγματικότητα στην Αλγερία. για λεπτό. Η ομάδα μου δεν προσυπογράφει το ψήφισμα. Εγώ όμως τη στηρίζω αυτή την πρόταση και κατά γράμμα και ως προς το πνεύμα. Πρέπει να είμαστε στο πλευρό των Αλγερινών Δημοκρατών που αγωνίζονται κατά τη διαφθορά, υπέρ τη θρησκευτική ελευθερία, τη κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, πράγματι υπάρχει καταστολή. Ε, υπάρχουν δημοσιογράφοι ε, και ε, αντιπολίτευση, αντιφρονούντε, οι οποίοι καταστέλλονται και σίγουρα δεν πρέπει να σιωπούμε. Λυπούμε που μόλις τώρα και όχι το Φεβρουάριο καταθέτουμε το ψήφισμα, γιατί τότε ήταν πολύ ισχυρό κίνημα αυτό το οποίο ξεσηκώθηκε και χρειαζόταν υποστήριξη Ξέρω ότι έχει ξεκινήσει εκλογική διαδικασία που είναι αμφισβητήσιμη και αμφισβητείται, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε εδώ για παρεμβάσεις ε, και να λέμε ότι ίσως είναι ξένοι πράκτορες ή διαδηλωτές. Υπάρχει αυτή η διαδηλωτέ, υπαρχει αυτη κατάσταση. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, αλλά ουσιαστικά είναι μια ε, υποστήριξη ακλόνητη που θέλουμε να παράσχουμε στους Αλγενούς, ιδίως στους νέους ε, που έχουν όρεξη για δικαιοσύνη, ανάγκη λαχτάρα για ελευθερία και δημοκρατία. Αυτό κάνουμε σήμερα, αυτούς υποστηρίζουμε. Έχει ο κύριος Πόσπισιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι θα υποστηρίξω την πρόταση ψηφίσματος. Είναι σαφές ότι θα πρέπει εμείς να προστατεύσουμε τους Αλγερινούς οι οποίοι εκφράζουν την επιθυμία τους για ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία. Και νομίζω ότι και ο διάδοχος της κυρίας Μογκερίνη έχει πολλά να κάνει ως προς αυτό. Πρέπει να γίνουν ελεύθερες προεδρικές εκλογές στην Αλγερία και επίσης θα πρέπει να πιστήσουμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στο θρησκευτικό μίσος που εκφράζει η πολιτική ηγεσία της χώρας ε, απέναντι στις θρησκευτικέ μειονότητες και δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στους χριστιανούς. Δυστυχώς οι εξελίξεις στην Αλγερία ε, δεν είναι καλές. All of Όλοι αυτοί θα πρέπει να παρετηθούν, φωνάζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες Αλγερινών απέναντι στους υπευθύνους της περίοδου Μπουτεφλίκα πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Γίνονται διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις τρεις μέρες την εβδομάδα και είναι όλο ένα και πιο ισχυρές. Και από την άλλη οι αρχές συλλαμβάνουν τους ειρηνικούς διαδηλωτές και τους βάζουν φυλακή με οκτώ μήνες μάλιστα ποινή. Πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να απελευθερώσει όλους τους ειρηνικούς διαδηλωτές. Ο στρατός είναι ο βασικός παίκτη στην ε, ζωή της χώρας και νομίζω ότι θα καθορίσει και το αποτέλεσμα των ε, εκλογικών αναμετρήσεων. Οι εκλογές ε, ε, δεν είναι μια υπόθεση δημοσίων σχέσεων και θα πρέπει να ελεγχθούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και να μην υπάρχει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας λογοκρισία όπως ακριβώς φαίνεται να ισχύει σήμερα. Κέλλη ένα λεπτό. Uh, Σας ευχαριστώ. Η Αλγερία είναι η γειτονική μας χώρα, πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις μαζί της, αλλά πρέπει ωστόσο για τον ίδιο λόγο να ανησυχούμε και για το τι συμβαίνει πρόσφατα, ειδικά το τι συμβαίνει με τις εκκλησίες. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και την ομάδα μου, γιατί είμαστε χριστιανοδημοκράτες και θέλουμε να υπερασπιστούμε τους χριστιανούς και τις χριστιανικές εκκλησίες ολόκληρο τον κόσμο. Δεν έχει νόημα να κλείνουν ε, οι εκκλησίες στην Αλγερία. γιατί ε, πρόκειται για αδικία. Πρέπει να πιέσουμε λοιπόν για να ε, σταματήσει αυτή η κατάσταση. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ε, διαδώσουμε την ειρήνη και την αγάπη στη χώρα και να επιμείνουμε για ελευθεροτυπία, ανεξιθρησκεία και ελεύθερες εκλογές και δίκαιες εκλογές κύριε πρόεδρε υπερασπίζομαι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου είτε χριστιανού είτε μουσουλμάνου να ασκεί το θρησκευτικό του καθήκον. ακόμα ένα ψήφισμα ακόμα μια φραστική καταδίκη για την αλγερία αν αυτά αληθεύουν που ακούσαμε και δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι δεν αληθεύουν ένα απλό ε, μια φραστική καταδίκη δεν βοηθά καθόλου νομίζω. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ω Κύπριο, ξέρω τι σημαίνει να σου στερούν το δικαίωμα να ασκήσει το θρησκευτικό σου καθήκον. Οι περισσότερε εκκλησίε στην Κύπρο, στα κατεχόμενα, έχουν μετατραπεί από του τούρκου σε στάβλου ακόμα και από και ρωτώ την κομισιόν πέρα από τη φραστική καταδίκη πέρα από τα ψηφίσματα θα λάβουμε μέτρα ω ευρωπαϊκή ένωση αν αυτό συμβαίνει στην αλγερία. ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Catch the Eye. Εξ ονόματο τη Επιτροπή, το λόγο έχει η κυρία Μογκερίνη. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie n'est pas seulement un pays voisin, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Αλγερία δεν είναι μόνο γείτονα, αλλά και εταίρο πολιτικός, οικονομικός. Είναι μια φίλη χώρα για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Η Αλγερία είναι και οικογένεια. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε χώρα λοιπόν, μεταξύ άλλων, αλλά για μια χώρα πολύ κοντινή μας, μια φίλη χώρα. για τον ε, αλγερινό λαό αισθανόμαστε νομίζω πρώτα απ' όλα εμείς οι Ευρωπαίοι ε, συγγένεια και φιλία. Νομίζω λοιπόν πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιβεβαιώσουμε ότι τους Αλγερινούς, οι Αλγερινοί μόνο μάλλον μπορούν να αποφασίσουν για το παρόν και το μέλλον της χώρας τους και ακριβώς γι' αυτό λόγο αυτό το λόγο οι Αλγερινοί πρέπει να είναι ελεύθεροι να εκφραστούν με τις εγγυήσει που προβλέπει το Σύνταγμά του και οι διεθνείς, συμφωνίε συμφωνίες, τις οποίες έχει υπογράψει η ίδια Αλγερία. Υπάρχουν κάποιες αρχές τις οποίες έχει συνυπογράψει η Αλγερία, κυρίως ε, αυτά περιλαμβάνονται στο Αλγερινό Σύνταγμα, αλλά και διεθνείς συμφωνίες, αλλά και με τη Συμφωνία Σύνδεσης που έχει η Αλγερία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνονται όλες οι θεμελιώδεις ελευθερίες και οι πολιτικές ελευθερίες. Ελευθερία έκφρασης, δικαίωμα στην ειρηνική συνέλευση, ε, στην ελευθεροτυπία, στις ελευθερίες που αγκιάται η δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι ακροχωνιαίος λήθος ε, του συντάγματος. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό όλοι οι Αλγερνοί να μπορούν να χαίρουν αυτών των δικαιωμάτων είναι ακριβώς αυτό το μήνυμα που διαρκώς διαβιβάζουμε στους αλγερινούς μας εταίρους και συνομιλητές σε όλα τα επίπεδα διαρκώς αυτούς τους μήνες και πιστεύω πως αυτό θα συνεχίσει να είναι το μήνυμα που θα συνεχίσει να στέλνει και η επόμενη Επιτροπή μόλις αναλάβει τα καθήκοντά της και θα συνεχίσει να το διαβιβάζει στους αλγερινούς συνομιλητές μας. Οι Αλγερινοί μπορούν να οικοδομήσουν συνένεση για το μέλλον της χώρας τους σύμφωνα με τις θεμητές προσδοκίες του λαού αυτό μόνο μπορεί να γίνει δημοκρατικά και ειρηνικά με σεβασμό στις αρχές και στις συμβάσεις που έχει υπογράψει η Αλγερία. Νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να έχει επαφές με όλους τους αλγερινούς φορείς όπως το έχουμε κάνει τόσα χρόνια ως γείτονες, εταίροι, φίλοι. Και νομίζω πως έτσι θα συνεχίσει και η επόμενη Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ε, έλαβα πέντε προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα. Η επόμενη συζήτηση αφορά την Κούβα και συγκεκριμένα την περίπτωση του Ζωζέ Ντανιέλ Φερέρ. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι υπάρχει δυνατότητα να υποβάλλετε έτοιμα για να σας δοθεί ο λόγος με τη διαδικασία του Catch the Eye ή τη διαδικασία της ερώτησης με γαλάζια κάρτα χρησιμοποιώντας τόσο τη συνήθη διαδικασία όσο και το ηλεκτρονικό σύστημα. Οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες και στην είσοδο του ημικυκλίου. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Λόπες Τζιλ για δύο λεπτά εκ των συντακτών. Me han hecho de todo mil torturas y violencia me han encadenado de Πολλά μου είπαν, με δέσανε χεροπόδαρα, με είχαν βάλει σε ένα κελί γεμάτο ε, κουνούπια, κρύο το πριν για 15 ημέρες. Ε, κινδυνεύει η ζωή μου. Αν δεν κάνετε κάτι θα πεθάνω. Τα έγραψε ο Χωσέ Δανιέλ Φερέρε σε μια επιστολή που κατάφερε να την περάσει από τη φυλακή και να φτάσει στη γυναίκα του. Και σήμερα ακούγονται αυτά τα λόγια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αφαιθεί ελεύθερο αυτός ο άνθρωπος που πάνω από 10 χρόνια τιμωρείται από τον καστρισμό επειδή προσπαθεί να υπερασπιστεί ανθρώπινα δικαιώματα. Η υπόθεση Φερέρ πραγματικά είναι αποτροπιαστική. Υπάρχουν όμως σαν αυτόν εκατοντάδες άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι ε, ε, συνείδηση ε, και πολλοί άλλοι που κρατούνται. Cuban Prisoners Defenders είναι η ομάδα που τεκμηριώνει την πραγματικότητα αυτών που λέω. Έχουμε πολιτικές διώξεις, ε, ε, δίμευση περιουσιών, φυλάκιση ε, συνηγόρων των μάλλον υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιφρονούντων. Αυτά συμβαίνουν σήμερα στην Κούβα. Θα πρέπει να απαιτήσουμε την άμεση απελευθέρωση του Χωσέ Ντανιέλ Φερέρ και όλων όσοι διώκονται στην Κούβα με βάση τη Συμφωνία για Πολιτικό Διάλογο και Συνεργασία ε, που έχει η Ένωση με την κουβανική κυβέρνηση. Μια συμφωνία που δεν είχε τελικά από ό,τι φαίνεται καμία θετική επίπτωση ε, για τον ε, πληθυσμό της Κούβας. Επίσης, πέραν του ψηφίσματος, θα ζητήσουμε για μια ακόμη φορά από την ύπατη εκπρόσωπο να λάβει υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διάλογο που έχει με τις κουβανικές αρχές και να ζητήσει να μπορέσει το Κοινοβούλιο μας να επισκεφθεί την Κούβα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τέρτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε να ψηφίσουμε εδώ μια πρόταση για τον Χωσέ Δανιέλ Φερέρ. Είναι ένας ε, πολιτικός ε, κρατούμενος, ένας από τους πολλούς ε, πολιτικούς κρατούμενους σε μια από τις πιο σκληρές δικτατορίες που υπάρχουν. Μια δικτατορία όμως με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο ο οποίος δεν τις αξίζει υπεγράφει διάλογος συνεργασίας αντίθετα με αυτούς οι οποίοι έλεγαν τότε ότι οι παραχωρήσεις προς μια δικτατορία η οποία δεν κάνει αυτή οι παραχωρήσεις που διώκει αυτούς που διαφωνούν, που επιμένει στο μοναδικό πολιτικό κόμμα και στην κομμουνιστική δικτατορία χωρίς καμία ελπίδα αλλαγής. Αυτή η μορφή συνεργασίας βοηθά την δικτατορία αυτή η οποία προσπάθησε μάλιστα να φανεί επεκτατικά στην υπόλοιπη Νότια Αμερική και βοήθησε στο να υπάρξει στη Βενεζουέλα την πιο πλούσια ίσως χώρα της ε, Λατινικής Αμερικής επέβαλε στη Βενεζουέλα λοιπόν ένα καθεστώς τρομοκρατίας και φόβου και αποτελεί απειλή για τις υπάρχουσες δημοκρατίες στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Σάντσες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έλεγα. Η σοσιαλιστική ομάδα έδειξε ε, ότι ανισχύει ιδιαίτερα για την υπόθεση Φερέρ και ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή του γιατί ξέρουμε ότι συνελήφθη αυθαίρετα ε, και δεν είναι αποδεκτές συνθήκες κρατησής του. Όμως δεν είμαστε υπέρ της ε, χειραγώγησης υπόθεση αυτής, ε, περιλαμβάνεται αυτό το θέμα στα κατεπήγοντα. Στο ψήφισμα όμως ουσιαστικά αυτό το οποίο τίθεται από αμφισβήτηση είναι το σχέδιο για το διάλογο και την συνεργασία δεν θέλουμε να γυρίσουμε ε, στο παρελθόν και στην παλιά ε, αμερικανική πολιτική που επιβάλλει κυρώσει σε ευρωπαϊκέ θέσει κτλ. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το νέο πλαίσιο, μπορούμε να ε, κάνουμε περισσότερα και να βοηθήσουμε για την περίπτωση Φερέρ και άλλων. Εμεί θέλουμε να έχουμε επαφή με την Κούβα. Βέβαια με κριτικό πνεύμα πάντα. Ευχαριστώ, κύριο Σπίν. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Ο... Πρόκειται για τον ε, υπηρέτη του κυρίου Τραμπ. γίνεται χειραγώγηση της δικαστικής διαδικασίας με κάθε εγγύηση ώστε ένας εγκληματίας που κατηγορείται για απαγωγή και που έχει χρησιμοποιήσει πιστόλι ενάντια στην γυναίκα του έγκυο 36 μηνών ε, δεν διώκεται στην Κούβα. Πολλέ, πολλές φορές ε, γίνεται ε, χειραγώγηση. Το ίδιο έχει γίνει και στη Χιλή και στη πραξικόπημα στη Βολιβία. Όλα αυτά μέσω του Αμερικανικού δακτύλου. Καθημερινά το βλέπουμε αυτό. Οι κατηγορίες ε, για την υποτιθέμενη επέμβαση της Κούβας σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι γελίες. Η μόνη παρέμβαση που κάνει η Κούβα σε άλλες χώρες και όχι μόνο της Λατινικής Αμερικής είναι με ε, ομάδες ε, μαέστρων και γιατρών. Θα πρέπει να το καταλάβετε. Η Κούβα υπάρχει θα πρέπει να στηρίξουμε μια σχέση ισότιμων με τον λαό της Κούβας. Το λόγο έχει η κυρία Χαραντσόβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χωσέλ Ντανιέλ Φερέρ ε, συνελήφθη αυθαίρετα. Θα πρέπει λοιπόν να ήταν ήδη ελεύθερος Σίγουρα εστιάζουμε στην υπόθεσή του σήμερα, όμω είναι ένα από τα πολυάριθμα παραδείγματα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να ε, συμβαίνουν ε, στην Κούβα. Είναι ένα από του 127 πολιτικού κρατουμένου, ο κ. Φερέρ. Ε, τόσοι είναι γνωστοί τουλάχιστον. Σε μια χώρα συμβαίνουν αυτά που έχει υπογράψει συμφωνίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται διατάξει του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υπεράσπιση τη δημοκρατία. Το 2017 ε, το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την προϋπόθεση στη συμφωνία αυτή να υπάρχουν ρήτρε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης όλων των κουβανών. Αυτό όμως δεν εφαρμόζεται ακόμα και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση απερίφραστα να πει ότι η Κούβα δεν τηρεί αυτή τη συμφωνία. Το πει ρητά η Ένωση και το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι να αναλάβουμε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση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 Η υπόθεση του Χωσέ Ντανιέλ Φερέρε δείχνει ξεκάθαρα ότι η κομμουνιστική Κούβα ποτέ δεν θα είναι σε θέση να ξεφορτωθεί το φορτίο του παρελθόντος της. δεν μπορεί να βασανίζει και να φυλακίζει τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τη δημοκρατία. Εγώ κατάφερα να συναντήσω τον ε, Χωσέ Ντανιέλ Φερέρ ε, στο Σαντιάκο της Κούβας και μάλιστα αρκετές φορές και σίγουρα δεν είναι τρομοκράτης όπως ε, ορισμένες δυνάμεις φιλοκουβανικές θέλουν να μας πείσουν εδώ στο Κοινοβούλιο. Αγαπάει τη χώρα του, θα πέθαινε για τη χώρα του ε, εκεί γεννήθηκε και εκεί θέλει να πεθάνει. Είναι ένας άνθρωπος που σέβεται όλους τους κανόνες που σεβόμαστε και εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα ήθελα να σας καλέσω, είπατε εκπρόσωπε, να χρησιμοποιήσετε τις επαφές σας και το κύριο σας ε, ως προς το κουβανικό καθεστώς και να πιέσετε για την άμεση του απελευθέρωση. Τρία αρένα για ένα λεπτό. Merci. José Daniel Ferrer se trouve aujourd'hui dans un état ο Ντανιέλ Φερέ βρίσκεται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση υγείας από την 1η Οκτωβρίου που συνελήφθη. Ε, υπέστη πολλά λόγω των πολιτικών του δράσεων, τις οποίες ασκεί ειρηνικά. Υπάρχουν άλλοι 120 ειρηνιστές δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι. Ο τελευταίος Πρόσφατα μάλλον ο Αρμάντο Σέσα Φορτούνη, ο οποίος μετά από 43 χρόνια στη φυλακή ε, έχασε πια τη ζωή του. Συνεπώς λοιπόν ο Χωσέ Ντανιέλ Φερέρ και όλοι οι φυλακισμένοι πρέπει να γνωρίζουν τους λόγους της κράτησής τους και να δικαστούν με σωστό δίκαιο και δημοκρατικό τρόπο. Οι αρχές της Κούβας λοιπόν θα πρέπει να πάψουν να διώκουν αυτούς που θέλουν να εκφράζουν τα αισθήματα ελευθερίας τους και να δώσει εγγυήσει η κυβέρνηση για την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της πολιτικής δραστηριότητας. Θυμίζω ότι έχει υπογράψει ε, ε, πολλές διεθνείς συμβάσεις η Κούβα ε, ανάμεσα σε αυτές και η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό τους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το, ε, τα σέβη μου κυρία Μογκερίνη. Το 2016 υπέγραψε μια συμφωνία η Ένωση με την Κούβα. Βασική της συνιστόσα είναι και προϋπόθεση ο σεβασμός της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων. Τον Ιούλιο του 2017 με ψήφισμά μας εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η ρήτρα αναστολή. Πάνω από 100 πολιτικοί κρατούμενοι και χιλιάδες αυθαίρετε σύλληψη σήμερα στην Κούβα. Δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση ο ο κύριος Φερέρ, αλλά δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι απολυταρχικό ε, κράτος η Κούβα ε, στο πλαίσιο της δυναστείας των Κάστρο. Δεν είναι απλά ένας τουριστικός ε, προορισμός, είναι ένα ε, στρατιωτικό καθεστώς. Ε, κρατάει ο Κάστρο Ραούλ, όπως και ο αδερφός του προηγουμένως, τα ενία της εξουσίας. Πρέπει να είμαστε συνεπείς τα άρθρα που δεν θέλουμε να τα εφαρμόσουμε, ας τα διαγράφουμε έχουμε από αυτές τις συμφωνίες. Γιατί και ο Κεβέδο έλεγε ότι το χρήμα είναι ο πιο ισχυρός ε, υπότης. Ευχαριστώ. Και δημοκρατίας, το λόγο έχει ο κύριος Ραήλ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ο Χωσέ Ντανιέλ Φερέρα ηγήθηκε του φιλιρινικού κινήματος ε, και ε, φαίνεται ότι κρατείται, εκτός μάλλον ότι κρατείται παράνομα, ε, βασανίζεται κιόλα. σε τέτοιες περιπτώσεις στην Καμπότζη, στην Ικαράγουα, στο Ιράν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δραστηριοποιηθεί πολύ πιο στεναρά και τώρα απλά κοιτάμε σαν να μην είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί μιλάμε για μια σοσιαλιστική δικτατορία δεν είναι τόσο ε, σημαντικό αυτό και επειδή είναι πολύ σημαντική για την ε, ισπανική οικονομία η χώρα αυτή και επειδή έχουμε ε, αλυσίδες ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις που ίσως τους το προτιμούν να είναι και έτσι κλειστή η Κούβα. Και μάλιστα έχουμε το Υπουργείο που στηρίζει την αυτή την κατάσταση. Όμως οι νόμοι και η δημοκρατία πρέπει να ισχύουν σε όλες τις χώρες. Ο κύριος Νικολάου Λαβάνος. Ο Χωσέ Ντανιέλ Φερέρ, που επιχειρείται με ψήφισμα να αεροποιήσετε, είναι επικεφαλή τη αποκαλούμενη Πατριωτική Ένωση τη Κούβα, δηλαδή τη πιο δραστήρια οργάνωση αντεπαναστατών στη χώρα. Συνελήφθη από τις κουβανικές αρχές μετά από καταγγελία πολίτη ότι μαζί με άλλου τρει ομοειδεάτε του τον ξυλοκόπησαν βαριά με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία. τα περί κακοποίησης ανεπαρκούς ποσότητας τροφής κτλ. είναι ψέματα που κατασκευάζει η κυβέρνηση των ηπα και η πρεσβεία του στην αβάνα με στόχο να εμφανίσει τα ανδρίκελά της σαν θύματα. ο φεραίρ εξάλλου είναι άλλος ένας περισσότερο αναγνωρίσιμος στα επιτελεία των ηνωμένων πολιτειών της αμερικής και της ευρωπαϊκής ένωσης παρά στη χώρα του και τον κουβανικό λαό. καταγγέλλουμε τη βιομηχανία ευρωενωσιακής σκοπής επιλεκτικής προστασίας δίθεν ακτιβιστών τις αλακάρτ υποκριτικές ανησυχίες της ευρωπαϊκής ένωσης περί καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποτελούν γνώριμο εργαλείο για την πιο αποτελεσματική διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε τρίτες χώρες ιδιαίτερα όταν αυτές οι χώρες δεν έχουν κυβερνήσεις της προτίμησης της ευρωπαϊκής ένωσης ή κρατών μελών της στο Έχουμε δυνατότητα. Τέσσερι συνάδελφοι που έχουν στήσει το Μπορούμε να του δώσουμε. Ε, ο κύριο Πόλτσακ, ε, καταρχά, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καταδικάσω ε, την σύλληψη και φυλάκιση του Χωσέ Δανιέλ Φερεργασία. Θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος. Οι κατηγορίες εις βάρος του δεν είναι σοβαρές. Θα πρέπει να ξεκινήσει ένας πραγματικός διάλογος με την κυβέρνηση της Κούβα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πρόκειται για μια ουσιαστική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν είναι μόνος του Φερέρ. Υπάρχουν άλλοι 120 πολιτικοί κρατούμενοι, οι οποίοι σαπίζουν ε, στις φυλακές της Κούβα. Θα πρέπει να καλέσουμε την κυβέρνηση της Κούβα να αλλάξει την κατάσταση. Εμείς στην Δημοκρατία της Τσεχίας βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε τα τελευταία χρόνια ε, τους ε, φυλακισμένους και τους πολιτικούς κρατούμενους στην Κούβα. Ο κύριος Γόλας, για ένα λεπτό ευχαριστώ πρόεδρε. Η Κούβα είναι λαμπρό παράδειγμα το ότι είναι δυνατό. Ε, ενάντια στα πάντα, ε, στις μεγάλες δυνάμεις που προσπαθούν ε, να ανατρέψουν την κυβέρνηση και να δολοφονήσουν τους ηγέτες άλλαξε το υποστηριζόμενο από τη CIA σύστημα. Υπάρχει τώρα ένα πρόγραμμα δράσης παρέχονται προμήθειες ε, στην Κούβα για να ουσιαστικά ε, δημιουργήσουν περισσότερη ε, φτώχεια, έλλειψη τροφίμων κτλ. Και τα καταφέρνουν από ό,τι φαίνεται πολύ καλά. είναι δεξιός ε, ε, με μακρύ ε, ιστορικό αυτός ο οποίος κρατείται. Δεν είναι όμως αυτό μόνο το θέμα. Το θέμα είναι να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις στην Κούβα για να μην υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Περέρα για να Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το ψήφισμα απαριθμεί ένα σωρό ψευδή στοιχεία που στόχο έχουν να δημιουργήσουν το πλαίσιο για να αιτιολογήσουν τις προτάσεις παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Κούβα και της αλλίωσης των αποφάσεων του λαού σε μια διεθνή προσπάθεια για καθοδήγηση του λαού της Κούβας είναι μία από τις πολλές προσπάθειες για να γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό έχει επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη που μάλιστα προτείνουν να ανασταλεί η Συμφωνία Συνεργασίας. Πρόκειται ε, Ωστόσο, δεν ε, ε, γίνεται λόγος για το εμπάργο που ισχύει εδώ και τόσα χρόνια κατά της ε, Κούβας, την επιδείνωσή του, παρά τις οικονομικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πρόοδου που έχει σημειώσει ο πρόοδος της Κούβας, ειδικά στον τομέα της υγείας, παρά το εμπάργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προχωρούμε. Κυρία Αντάλη για ένα λεπτό. Ντέιλι, μάλλον. Thank you, um, President. I would like to... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα εγώ να εκφράσω την ε, αντίθεσή μου με το περιεχόμενο και το ύφος αυτής της απαράδεκτης πρότασης. Έχει σαν στόχο την απομόνωση του λαού της Κούβα και της κυβέρνησής της, υπακούοντας τις Ηνωμένε Πολιτείες και εντασσόμεθα και εμείς πλέον σε μια επιθετική στάση απέναντι σε αυτόν τον τόσο ανθεκτικό λαό. Το περιεχόμενο έτσι και αλλιώ είναι λανθασμένο. Ο Φερέρ είναι ένας τραμπούκος πολιτικός δίκαια φυλακισμένος. Ε, και φυσικά οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αυτές οι οποίες τον υπερασπίζονται και υπερασπίζεται φυσικά και την παρέμβαση ε, των Αμερικανών και αν δεν υπήρχε η ανθρωπιστική βοήθεια την οποία έδιδε η Κούβα ε, στη Βολιβία, στη Βενεζουέλα και σε άλλες χώρες η κατάσταση θα ήταν πάρα πολύ κακή. Και εμείς ε, συγχαίρουμε την κυβέρνηση της Κούβα για τη στάση της. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνω τη συζήτηση με την κυρία Μογκερίνη που θα κλείσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο Σεντανίλ Φέρερ από την Πατριωτική Ένωση της Κούβα, συγέτης, 1η Οκτωβρίου συνελήφθη ε, στο σπίτι του, στο Σαντιάγο Δε Κούβα. Κρατείται εκτοτε περιορισμένες επισκέψεις, από την οικογένειά του έχει δεχθεί, η υγεία του είναι εύθραυστη, έχουμε αναφέρει την υπόθεση και αυτή αλλά και άλλων ε, κρατουμένων ε, στις κουβανικές αρχές και στην Αβάνα και στις Βρυξέλλες και πιο πρόσφατα σε επίπεδο επικεφαλής αντιπροσωπιών. Και να Νοεμβρίου πιο πρόσφατα με το Υπουργείο Εξωτερικών. Σήμερα η ε, γονείς του, μάλλον η οικογένειά του ε, και τα παιδιά του τον επισκέφτηκαν μετά τη δική μας παρέμβαση. Πολλές φορές έχουμε πει ότι περιμένουμε η Κούβα να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όλων των πολιτών και το δικαίωμα σε δικαιή δίκη. Πάντοτε αναφέρουμε και προβάλλουμε τέτοιες υποθέσεις αυτού του κυρίου Φερέρ. Συντονισμένα με τα κρατημέλη και εκ των προτέρων ε, προσπαθώντας ε, να έχουμε ένα ανοιχτό ειλικρινή διάλογο με την Κούβα. Δεν έχουμε ταμπού σε όλα τα επίπεδα θέτουμε αυτά τα ζητήματα, όποτε αυτό το κρίνουμε απαραίτητο. Και δυστυχώς αυτό γίνεται πολύ συχνά. Δεν συμφωνούμε απόλυτα σε όλα με την Κούβα. Ακριβώς γι' αυτό έχουμε αυτό το διάλογο, επειδή δεν συμφωνούμε σε όλα μεταξύ μας. Και είμαι υπερήφανη που έχει πλέον ανοίξει μια νέα σελίδα και μια νέα φάση στη σχέση μας με αυτή τη χώρα. Με την πλήρη υποστήριξη, το τονίζω αυτό, όλων των κρατών μελών. Μηδενός εξαιρουμένου ανεξαρτήτως και της ε, πολιτικής ε, κατεύθυνσης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδες μέρος αυτής της συμφωνίας και έχουμε επαφή με την κουβανική ηγεσία και με κριτικό πνεύμα. Εκφράζουμε και τις διαφωνίες μας και ζητούμε κάτι να γίνει για τα κακοσκήμενα Και ακριβώς ε, αντικείμενο του πρόσφατου διαλόγου που είχαμε με την Κούβα ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Μόνο αν είναι πλήρως σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν υπάρχει χώρος για την κοινότητα των πολιτών μπορεί να υπάρξει και οικονομική ανάπτυξη η οποία να είναι βιώσιμη. Έτσι μπορούμε να συνοδεύσουμε τη χώρα στην πορεία της προς τον εξυγχρονισμό. Είναι και ένας από τους στόχους της συμφωνίας μας. Να πλαισιώσουμε τη χώρα που μεταρρυθμίζει το πολιτικό-οικονομικό της μοντέλο και δημιουργεί μια, οικοδομή, μια οικονομία σε πιο σταθερά θεμέλια όπου όλοι μπορούν να έχουν επίσης τις ίδιες ελευθερίες αλλά και τα ίδια δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο της μεσεδιάταξης και πρωτού προχωρήσουμε στην ε, επόμενη συζήτηση για την ΑΕΤ. θα ήθελα να σας πω ότι ο πρόεδρος ομάδας ε, του ΕΛΚΑ μας ε, έδωσε την εξής, τις εξής αλλαγές σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος ο κύριος Μοντρεάνου αντικαθιστά τον κύριο Μπουσόη και με τη σειρά του ο κύριος ε, Μπουσόη αντικαθιστά την κυρία Βάλεάν στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Οι αποφάσεις αυτές ε, αρχίζουν να ισχύουν από τώρα. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι IT και θέλω να σας πω ότι μπορείτε για τις μπλε κάρτες και για την διαδικασία Catch να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σύστημα. Εδώ λοιπόν ξεκινά η συζήτηση για την IT με πρώτο ομιλητή, ε, το συντάκτη, ε, μεταξύ άλλων ο κ. Δεχόφσκι. Είπατε εκπρόσωπε. Ε, ε, η ΑΕΤ εδώ και χρόνια είναι πολιτικά σταθής. Είναι μια χώρα όπου επικρατεί μεγάλος βαθμός διαφθοράς, όπου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου δημοσιογράφοι χάνουν τη ζωή τους. Είναι μια χώρα όπου οι ατομικές ελευθερίες είναι περιορισμένες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει την ικανότητά της να ε, κάνει διάλογο, να διευκολύνει το διάλογο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξει η κατάσταση στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν που μετά το σεισμό βοήθησε στην αποκατάσταση αυτής της όμορφης χώρας. Όμως θα πρέπει να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση του πολιτικού κλίματος στην κοινωνία της ΑΕΤΗΣ. Αυτό είναι ένα από τα χειρότερα στη πλανήτη. Το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους στοχούς δεν είναι το χειρότερο στη χώρα. Το χειρότερο είναι η αστάθεια και η και η αδυναμία πρόβλεψης. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα πέσει θύμα ενός εγκλήματος ή μιας πολιτικά κινούμενης βίας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει στη χώρα. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ουρτασούν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ γιατί είναι μία από τις ε, χώρες που είναι η μεγάλη ξεχασμένη. Είναι μια πολύ φτωχή χώρα με αναπτυξιακούς δείκτες ε, υπό το μηδέν. Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες αναπτυξιακους δεικτες υπο το μηδεν αυτο που συμβαινει το τελευταιες μερες μας υποχρεώνει να καταδικάσουμε τη βία, την καταστολή. Εγώ έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες ότι ο πρόεδρος Μωής που τον κατηγορούν οι διαδηλωτές για διαφθορά και υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μάλλον είναι αλήθεια. Ε, λοιπόν θα πρέπει ίσω να γίνουν εθνοεκλογές για να αποκατασταθεί μια κάποια τάξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίζει, πιστεύω, με τα μέσα από συνεργασίε που έχει. Πάντως είναι προφανές ότι ενώπιον των θεσμικών και των ε, θεσμικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα πρέπει να είναι δύσκολο να σταλεί και η βοήθεια και η στήριξη. Άρα λοιπόν η στήριξη στον εθνικό διάλογο θα πρέπει να έχει προτεραιότητα κατά τώρα και με τα πέντε δευτερόλεπτα που μου μένουν επειδή τελευταία φορά σας βλέπουμε είπατε εκπρόσωποι εδώ να σας ε, ευχαριστήσω και να σας για τη δουλειά και τη συνεργασία τα τελευταία πέντε χρόνια τις δραστηριότητες, πρωτοβουλίες που αναλάβατε τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Τσαρνέτσκι είναι ο επόμενο ε, συντάκτη, Για ένα λεπτό. Ε, ε, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μογκερίνη για τα πέντε χρόνια αυτά συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσωπικά εγώ συνεργάστηκα μαζί της σε σχέση με την πολιτική γειτονίας. Νομίζω ότι η συνεργασία ήταν αρκετά αποτελεσματική. Η ΑΙΤ είναι μία από τις φτωχότερες βέβαια χώρες στον κόσμο. Πρόκειται για μία χώρα η οποία έχει να αντιμετωπίσει κύκλι... κλιματολογικές καταστροφές, φυσικές καταστροφές. Ανθρωπιστική βοήθεια δίδεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συγκεκριμένη χώρα και η ανθρωπιστική βοήθεια αυτή δεν ελέγχεται πλήρως και δεν φτάνει πάρα πολύ συχνά στους τελικούς παραλήπτες. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τη βοήθεια αυτή πάρα πολύ κοντά. Να δούμε ακριβώς πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα τα οποία δίδονται. Η Πολωνία είχε στείλει <clears throat> μια ομάδα στρατιωτική στην, στην για να βοηθήσει. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ζωρίνιο. Κυρία Είπατε εκπρόσωπε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας ε, για την εξαιρετική θητεία που μόλις ε, ολοκληρώσατε. Η πολιτική κατάσταση και η κοινωνική κατάσταση στην ΑΕΤ είναι αβάσταχτη. Οι διαμαρτυρίες στους δρόμους είναι ένα αιτιολογημένο μήνυμα ε, αντίδραση ενάντια σε μια τέτοια διοίκηση και ενάντια σε ζωή, ζωής πραγματικά απέσιε. Η ε, δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστεί με το λαό στην πορεία της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της δημοκρατίας, σε σεβόμενη το κράτος δικαίου, πρέπει να υπογραμμιστεί και να εφαρμόζεται μόνιμα. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου που σήμερα συζητάμε θα πρέπει να ε, καταδικάσει αυθυρότατα τη βία ο απέναντι στην στην ελευθερία λόγου στην ΑΕΤΗ είναι σημαντικό οι διεθνεί οργανισμοί να αυξήσουν την προσπάθεια για ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά βέβαια όλα αυτά δεν θα έχουν την απαραίτητο αντίκτυπο εάν το ίδιες, οι ίδιε οι αρχέ τη ΑΕΤ δεν εγγυηθούν άμεσα την ελευθερία έκφραση και το σεβασμό των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ε, μεταξύ των συντακτών και αυτό ο κύριο Ουρμπάν Κρέσπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε γιατί είναι η φτωχότερη χώρα της Αμερικανικής Υπήρου, είναι θύμα των πολιτικών των ε, διεθνών οργανισμών με τεράστιο χρέος και με εθνούσα τάξη που ουσιαστικά γεμίζει τις τσέπες της με χρήματα. Και ο λαός καταδικασμένος στην εξαθλίωση. Αυτή είναι η ε, συνταγή του καπιταλισμού, του καζίνο. Πρέπει να πάψει η νεοφιλελεύθερη πολιτική. Έχουμε δολοφονίες από την αστυνομία που φαίνεται να συνδέεται με εγκληματικέ οργανώσεις και ε, έχουν φαίνεται κακοποίηση επίσης ε, και σεξουαλικά πολλές γυναίκες. Δεν θα πρέπει να υπάρχει συνένοχη σιωπή από τη διεθνή κοινότητα. Θέλουμε οι πολιτικές λιτότητες ε, να πάψουν να μπορούν οι Αιτιανοί να αντιμετωπίζουν το μέλλον τους με αξιοπρέπεια. Ελπίζω να μην χρειαστεί ε, να, σας, ε, να μας λείψετε πάρα πολύ με αυτό που έρχεται ε, για μας την επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε με την κυρία Χόβεβα, εκ μέρους των συντακτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι έχουμε να κάνουμε με μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Μία χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από βία, ε, διαφθορά, σύγχρονες μορφές ε, ε, σκλαβιάς Πραγματικά είναι μια χώρα στα έλεγα στην άκρη του χάους πια. Δεν υπάρχει συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, υπάρχει πρόβλημα στον τομέα της διατροφής, υπάρχει τρομακτική ε, χρήση βίας, δεν υπάρχουν κατεπίγουσες ιατρικές υπηρεσίες, ε, η εκπαίδευση δεν λειτουργεί. Λοιπόν, γι' αυτό απαιτούμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να σταματήσουν πλέον να ασκούν βία, να σταματήσουν να δημιουργούν προβλήματα στην ζωή των πολιτών τους και να σταματήσουν τις δολοφονίες των δημοσιογράφων. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στη συζήτηση ε, με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Παρακολουθεί ο κύριος Κέλλη. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πράγματι την Αϊτή μπορούμε να την περιγράψουμε σαν μία από τις ε, ανήθικες χώρες του κόσμου μέσα σε όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει ουσιαστικά ε, βουλή, υπάρχουν ε, πολλαπλές μορφές βίας βάρος του πληθυσμού Υπάρχουν φυσικά διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, των κοινοτήτων ΛΟΑΤΒ. Γενικά υπάρχουν τρομακτικές καταστάσεις και σε επίπεδο οικογενειακής ζωής και δυστυχώς τα παιδιά σύν της άλλης και κυρίως δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, δεν υπάρχει ουσιαστικά εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τουλάχιστον αυτό να το διασφαλίσουμε. Δεν μπορεί να υπάρχουν παιδιά τα οποία να μην έχουν την δυνατότητα να μορφωθούν. ευχαριστώ, πολύ. Νίνα Τζίλ από τους και Δημοκράτες είναι επόμενη στον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη όπως ακούσατε ήδη η IT βρίσκεται ε, ένα βήμα πριν από την καταστροφή. Πυροσβολισμοί, ε, τουλάχιστον 20 άτομα έχουν δολοφονηθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας και δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό, δεν υπάρχει πρόβλημα στον τομέα, υπάρχει μάλλον σοβαρό πρόβλημα στον τομέα της ενέργειας και φυσικά το σύστημα υγείας είναι κατεστραμμένο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια λύση η οποία ε, να δώσει ε, και κάποιες εναλλακτικές στο πρόβλημα της διαφθοράς η φόρος ανάπτυξη της νήσου αυτής ε, είναι απαραίτητη αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την διαφθορά. Τι μοχλούς χρησιμοποιείται, γιατί εμείς μέσα από το EDF δίνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια βοήθειας και παρόλα αυτά δεν έχουμε ελαφρύνει τα προβλήματά τους. Θέλω επίσης κυρία Μογκερίνη να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και να ευχηθώ ότι καλύτερο στο μέλλον. Συνεχίζουμε. Επόμενη είναι η κυρία Ροντρίγκε Ράμο, εκ μέρου τη ομάδα Renew Europe. Μόνιμη ανθρωπιστική κρίση στην Αϊτή, μια χώρα που ναι ε, έχει ε, περάσει την ε, κρίση της φυσικής καταστροφής και βιώνει άλλες κρίσεις, ανθρωπιστική, τομέα τα κτλ. Επίσης πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, ανασφάλεια και δυστυχώς διαφθορά. 38.000 άνθρωποι από το σεισμό του 2010 παραμένουν άστεγοι και από το Σεπτέμβριο υπάρχει μια βίαιη κατάσταση, πολύ ανησυχητική, ακριβώς λόγω των διαδηλώσεων της κοινωνίας κατά της κυβέρνησης και της έλλειψης ε, εφοδιασμού. Ε, κατάσταση αυτή ε, επιδεινώνεται με 40 θανάτους, τρεις δολοφονίες δημοσιογράφων που κάλυπταν ακριβώς ε, τις ε, ταραχές αυτές και νομίζω ότι πρέπει να στήσουμε την πάυση της βίας. Θέλουμε μια πολιτική λύση μέσω δίκαιων εκλογών και βέβαια ανθρωπιστική βοήθεια σε μια χώρα που το 40% του πληθυσμού εξαρτάται από τη διεθνή επιστηστική βοήθεια. Ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία κυρία Επίτροπε. Πρώτα, ευχαριστώ πολύ. Επόμενη στη συζήτηση ε, από τους μη εγγεγραμμένους η κυρία Αντινόλφη. Η κατάσταση στην Αϊτή συνίσταται από βία, από διαφορά, από φτώχεια από σοβαρά προβλήματα γενικότερα και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει μεγάλη αξία, δεν μπορούμε να κοιτάμε χωρίς να παρέμβουμε. Ε, τα χιλιάδες παιδιά που πολλούνται στην Αϊτή ως οικιακή βοηθή από τις φτωχές οικογένειες. Δεν ε, υπάρχει δικαιοσύνη. Φυσικά είναι επιστημονική φαντασία η ισότητα των φύλων και σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία μας έχει δώσει η Επίτροπος για τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα ε, στην ε, IT έχασαν τη ζωή τους τον προηγούμενο μήνα δεκάδες άνθρωποι σε συγκρούσεις ένοπλες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τα επιτρέπουμε όλα αυτά. Γιατί τα επιτρέπουμε. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Μογκερίνη για την παρουσία της τα τελευταία χρόνια και της εύχομαι ό,τι καλύτερο για την περαιτέρω σταδιοδρομία της. Ευχαριστούμε και τώρα ο συνάδελφος Καστάλτο δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Α, όχι, εδώ είστε, παρακαλώ. Βιαστείτε γιατί περιμένουμε. Ανοίξτε το μικροφωνό σας. You can use every mic you want, but just stop, please. <laughs> Όποιο μικρόφωνο σας βολεύει. Do you want me to continue with... Θέλετε να συνεχίσω με το Catch the Eye καλύτερα. Ναι. Οπότε περνάμε στους συνεδάλφους που έχουν ζητήσει το λόγο βάσει της διαδικασίας Κατσδιάη. Ξεκινάμε με τον κύριο Πασάλτζιλ από το ΕΛΚ. Πόσπισιλ, με συγχωρείτε, το διάβασα λάθος. Θέμα γραφικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τελικά κατάλαβα ότι πρόκειται για μένα. Πολύ σύντομα ήθελα να υποστηρίξω το ψήφισμα για την ΑΕΤ, διότι στην προηγούμενη ιδίω στην προεκλογική περίοδο, ε, μιλήσαμε για την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη χώρα αυτή που είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Τελευταία είδαμε οι εντάσει να κλιμακώνονται, ο κόσμο να κατεβαίνει στου δρόμου για να διαδηλώσει και να διαμαρτυρηθεί κατά τη ε, επιδείνωση του βιωτικού του επίπεδου. Είναι πολλοί που βρίσκονται στη γραμμή του επίπεδου τη φτώχεια. Υπάρχει παιδική δουλεία, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι νέοι τη εκπρόσωποι, να προσπαθήσουν να οργανώσουν διάλογο με τη χώρα αυτή. Κάτι που να οδηγήσει τουλάχιστον στην ε, διαμαρτυρία των πολιτών ελεύθερα χωρίς να διώκονται. Θα πρέπει η κυβέρνηση στην ΑΕΤ να κοιτάξει να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των πλέον φτωχών της χώρας. Δεν πρέπει να αδιαφορούμε για το γεγονός ότι και στην ΑΕΤ τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται. Ευχαριστούμε. Τσουχοντάρου. Danach. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μογγυρίνη, σας ευχαριστούμε γιατί ε, στη διαδρομή που κάνατε στη θητεία σας αντιμετωπίσατε ένα σωρό πυρκαγιές τις οποίες καταφέρατε όλες να τις σβήσετε και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε να έχετε επιτυχίες. Πάντως ήρθε η ώρα το Κοινοβούλιο και εμείς οι βουλευτές να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο διεθνή ε, με διαφάνεια για να μπορέσουμε να παρακολουθούμε τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη αυτούς που τα καταπατούν γιατί θα πρέπει όλοι μαζί να βρούμε λύσεις. Και πάλι συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε. Κύριε Καστάλτο, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρώτα πρώτα, ευχαριστώ για την κατανόηση. Έχουμε αυτέ τι ε, διαμαρτυρίε που θέλουν ο Μόζε να παραιτηθεί. Αυτό έχει ξεκίνησε από τον Ιούλιο. Είναι μια επανάσταση του λαού που ξεκίνησε ε, από τότε που ακυρώθηκαν οι επιδοτήσει από την κυβέρνηση για τα καύσιμα και έχουμε το Δούνο του που βοηθάει να ξεκίνησε η χώρα και όλα αυτά ε, φέρνουν τρομερές συνέπειες για τη χώρα, μεγάλες δυσκολίες επιπλέον από το εμπάρκο που υπάρχουν ε, από τη ΣΥΠΑ στην Βενεζουέλα. Δύσκολο να φανταστούμε τι γίνεται γιατί είναι η πιο ε, φτωχή χώρα του Δυτικού Ημισφαιρίου και πρέπει να γίνουν κάποιες αντισταθμίσεις για να προστατεύσουν τους πιο φτωχούς της κοινωνίας. Όμως τώρα θα πρέπει να εγκαταλείψει την ε, Προεδρία και αυτές του τις ε, πολιτικές έχει τη στήριξη ε, των ΙΠΑ και του ομίλου των φίλων της ΑΕΤΗΣ που είναι Ευρωπαίοι. Κάπως πρέπει να γίνει για να υπάρξει για τους φίλους Αιτιανούς δημοκρατία, δικαιοσύνη και ισότητα. Πόλτσακ, ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και να αρχίσω με το πώς έχει η κατάσταση. Τι έχουμε, έχουμε ένα πλήθος και πυροβολισμού στον αέρα. Αυτό δείχνει την εικόνα της ακραίας φτώχειας στην χώρα. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι να καταδικάσουμε τα όσα γίνονται εκεί. Βία και εξεγέρσεις γίνονται κατά της ε, διεφθαρμένης και κατά του Προέδρου. Τα θέματα είναι η αύξηση της τιμής καυσίμων και φαγητών, κλιμάκωση των πραγμάτων, φόνος δημοσιογράφου ε, πρόσφατα και στην κατάταξη ε, των χωρών με κίνδυνο για τους δημοσιογράφους γιατί ε, δεν τα πάει και πολύ καλά, κατρακυλάει, άρα θα πρέπει να γίνει διερεύνηση ε, της διαφθοράς και επίσης να καλυφθούν οι ανάγκες του κόσμου σε φαγητό οπότε θα πρέπει η ύπατη εκπρόσωπος ε, επίσης να έχει επιτυχία και συνέχεια της διαδρομής της και την ευχαριστούμε για όσα έκανε. Ε, τώρα θα δώσουμε το λόγο στους βουλευτές. Ε, κύριε Γουόρτ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και στο τέλος θα πάρει το λόγο η κυρία Μαγκερίνη. Uh, thank you very much, President. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουν ξεσπάσει αυτές οι διαμαρτυρίες και λόγω της έλλειψης ε, καυσίμων, βία και ε, στρατεία κατά του Προέδρου και σύμφωνα με τον ΟΗΕ υπάρχουν τα εξής στοιχεία. Τουλάχιστον 42 είναι οι νεκροί και πάρα πολλοί οι τραυματίες κατά αυτές τις διαδηλώσεις ε, ανασφάλεια, βία, ήδη τα πράγματα ήταν ε, κακά, γίναν χειρότερα, ε, ανισότητα, διαφθορά, πάνω από το ένα στους τρεις στην ΑΕΤ χρειάζονται βοήθεια γιατί δεν έχουν να φάνε τα βασικά. Μιλάμε για 7 εκατομμύρια που πεινάνε, θα πρέπει ο ΙΕ να βοηθήσει, θα συνεργαστεί με τις αρχές της χώρας για κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια άλλο θλιβερό το οποίο έγινε και είναι ε, δύο είναι το τι γίνεται κατά των γυναικών στις κρατικές φυλακές. Οι γυναίκες βιάζονται γιατί είναι στα ίδια κελιά με τους άντρες. Είπαμε ότι έχουμε αυτέ τι 16 ημέρε δράση για να σταματήσει βία κατά των γυναικών. Οπότε προσπαθήσουμε για αυτέ τι γυναίκε σε μία από πιο φτωχέ χώρε του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφε. Για να κλείσει τη συζήτηση, το λόγο έχει η κυρία Μογκερίνη. Παρακαλώ. Η χώρα αυτή της Αμερικής όπως και άλλες έχει κρίση πολιτική, οικονομική και κοινωνική. Ο πληθυσμό διαμαρτύρεται κατά του τρόπου διακυβέρνηση τη χώρα αυτή τη στιγμή, κυρίω κατά τη διαφθορά και του τρόπου που διαχειρίζονται την κρίση με υψηλού αριθμού ε, φτώχεια. Οι νέοι, οι ε, γεωργοί και κτηνοτρόφοι είναι ε, στην πρωτοπορία των ε, διαμαρτυριών ε, και είναι συνταγματική η κρίση στη χώρα χωρίς Βουλή και κυβέρνηση που να μπορεί να κρατήσει τα ενία. Πολλοί από εσά αναφέρατε τις ελλείψεις που παραλύουν τη χώρα από το καλοκαίρι. Ε, σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικοί θεσμοί, ε, δημόσιες υπηρεσίες και μεταφορές στη χώρα δεν προσφέρονται συστηματικά. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι απαραίτητη και η χώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Οι πολιτικέ ε, τοποθετήσει και ιδεολογίε γίνονται όλο και πιο ριζοσπαστικέ και η βία αυξάνεται και διωγγώνεται. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις της ε, παρούσας κρίσης σε συνδυασμό με τη, σε συνεργασία με τους θεσμούς του ΟΗΕ φροντίζοντα να κάνουμε τις ανάλογες έρευνες και ανακρίσεις για τα ε, εγκλήματα που διαπράττονται. Θα πρέπει να μπορούν να διαμαρτύρονται οι πολίτε ειρηνικά και χωρίς προβλήματα και να αποφεύγονται οι βίες ενέργειε. Το λέω και το είπα και στις αρχές του μήνα εκ μέρους των 28 κρατών μελών και θα κοιτάξουμε να οργανώσουμε εθνικό διάλογο με την ΑΕΤ για να βρούμε εάν μπορεί να υπάρξει λύση συνένεση στην κρίση αυτή, που είναι πολιτική, οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει και με άλλους δωρητές την προσφορά άμεσης βοήθειας για την ανακούφιση της κατάστασης εντός της χώρας, γιατί οι ανθρωπιστικές, συνθήκες είναι δραματικές. Δεν μπορούν να κρατήσουν τα πράγματα έτσι, όχι μόνο από ανθρωπιστική σκοπιά, αλλά και λόγω της πολιτικής διαδικασίας που πρέπει να γίνουν ευνοϊκές, ε, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτή η χώρα. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου ολοκληρώνοντας Καταρχάς να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, κάτι που έχω κάνει σπάνια σε αυτό το ημικύκλιο τα περασμένα χρόνια. Να σας ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Η αρχή της κοινοβουλευτικής αυτής θητείας, οι τελευταίοι μήνες για μένα, ε, έδειξαν ότι οι βουλευτές που βρίσκονταν στα έδρανα αυτά, όπως και οι προκάτοχοί τους, ήταν πάντοτε ε, θετική στη συνεργασία μας. Έδιναν πάντα μεγάλη σημασία στο ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου λοιπόν είναι θεμελιώδης όχι μόνο για την δημοκρατία στην Ευρώπη, αλλά και για την δουλειά μας για την ειρήνη την ασφάλεια, για μια εξωτερική πολιτική που να βασίζεται στην συνεργασία όλων στον κόσμο, στο σημερινό κόσμο ιδίω. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλους στο Κοινοβούλιο, τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους του, όλε τι πολιτικέ ομάδε και όλο ιδιαίτερο τι δύο κοινοβουλευτικέ επιτροπέ με τι οποίε συνεργαζόμουν ε, στενότερα, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ανάπτυξη, οι, πάντοτε, οι οποίε πάντοτε στήριζαν ουσιαστικά τη δουλειά μου τα τελευταία χρόνια. Χίλια ευχαριστώ. Äh, κυρία Επατεκπρόσωπε, κυρία Μογκερίνη, νομίζω ότι μπορώ να πω και εξ ονόματος ε, του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ότι σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας με το Κοινοβούλιο και τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και για την προσωπική σας ε, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα, στη συνεργασία ε, των πολυμερών θεσμών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ειλικρινά για την εργασία σας και για το πάθος το οποίο σας χαρακτηρίζει και έχετε επιδείξει. Ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση έχουν κατατεθεί έξι προτάσεις ψηφίσματος ε, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και διακόπτω τη συνεδρίαση μέχρι τις 11.30 οπότε θα ακολουθήσουν και οι ψηφοφορίες.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 Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και βουλευτές, καθίστε για να αρχίσουν οι ψηφοφορίες. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Σας παρακαλώ, καθίστε. it's θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους 500 εκατομμυρίων πολιτών στην σημερινή Ολομέλεια. Θα ήθελα να αρχίσω με μια ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού 2018 ε, κάθετος 1725 ε, του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου του 2018 η διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της σήμερα και μετά τις συνομιλίες στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ενέκρινε το το κοινό διορισμό Κοινοβουλίου και Συμβουλίου του κυρίου Βόιτσε Κράφαλ Βιαβορόφσκι ε, στη θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο Πρόεδρος θα υπογράψει την απόφαση διορισμού ε, μαζί με τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Μπορούμε να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Κύριε Βέμπερ, έχετε διαδικαστικό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σιωπά σε σχέση με τα τεκτενόμενα αυτή τη στιγμή στη Μάλτα γύρω από τις έρευνες που διεξάγονται για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Δάφνη Καρουάνα Γκαλίσια και σίγουρα το κοινοβούλιο μας δεν μπορεί να σιωπά και η αίθουσα τύπου φέρει το όνομά της. Αυτή την ε, εβδομάδα δύο υπουργοί παρετήθηκαν όπως και ο προσωπάρχης του ιδιαίτερου γραφείου του κυρίου Μουσκάτου, πρωθυπουργού υπό το φως των νέων αποκαλύψεων. Όλοι αυτοί εμπλέκονται ε, στις έρευνες της Δάφνη ε, Καρουάνα Γαλήσια πριν δολοφονηθεί. Τους έχει προστατεύσει όμως όλο αυτό τον χρόνο ο Πρωθυπουργός Μουσκάτ με βίες και σφοδρές επιθέσεις ε, κατά ε, όσων τους κατηγορούσαν. Η κατάσταση στη Μάλτα έχει συνέπειες για όλο το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει τώρα, περισσότερο από ποτέ, να καταστήσει σαφές στις αρχές της χώρας ότι ε, όταν υπάρχουν πολιτικές δολοφονίες δημοσιογράφων θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες συνέπειες. Έχω ακούσει το Κοινοβούλιο να διατρανώνει τις απαιτήσει του για την ελευθερία του τύπου και το κράτος δικαίου σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Σήμερα πρόκειται για τη Μάλτα. Ας υψώσουμε από κοινού τη φωνή μας όλοι μαζί. Η Ράτσε Γκαρσία Πέρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ανέκαθεν ήταν, είναι και θα είναι το κράτος δικαίου. Ανέκαθεν. Δεν επιλέγουμε πρόσωπα όταν μας συμφέρει, όταν σταματάει να μας συμφέρει. Θέλω να πω όμως το εξής. Το κράτος δικαίου λειτουργεί όταν συλλαμβάνονται οι υποπτοί και κινούνται οι ε, δικαστικές διαδικασίες. Αυτό συνέβη την περασμένη εβδομάδα στη Μάλτα. Συνελήφθη ένας ύποπτο και ακολουθεί η δικαιοσύνη το δρόμο της. Το κοινοβούλιο μας θα πρέπει να σέβεται ε, τις δικαστικές διαδικασίες και να μην επεμβαίνει σε αυτές. Θέλω πάντως να διευκρινίσω ότι η ομάδα μας ανέκαθεν είναι με το μέρος της αλήθειας και τη δικαιοσύνης. Άλλοι είναι εκείνοι που θα πρέπει να ξέρουν και να καταλαβαίνουν ε, ότι δεν είναι αυτά κατ' επιλογή τα πράγματα και νόνοι το. Και δεν πρόκειται να σταματήσω. Δεν πρόκειται να σιωπήσω. Μπορεί αυτό να σας ενοχλεί που διευκρινίζω εδώ αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη δεν είναι επιλεκτική. Και εμείς ε, δεσμευόμαστε από τα λόγια μας και από τα έργα μας και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ελπίζω την επόμενη πενταετία πάντα να είναι με το κράτος δικαίου, όπου και αν είναι αυτό, σε οποιαδήποτε χώρα και με οποιαδήποτε κυβέρνηση. And now we should proceed. Ωραία. Προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ, έχετε τις κάρτες σας, ετοιμαστείτε. Διαδικαστικό. Ποιο. Yeah. Πρόεδρε, ο κύριος Γκίγκολτ, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι αυτό που είναι κρίσιμο για την κατάσταση στη Μάλτα είναι κατεπηγόντως να στείλουμε επιτροπή εξεταστική των πραγμάτων, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο Βέμπερ για αυτά που λέει. Θα πρέπει να δούμε αυτά που έχει αποφασίσει το προηγούμενο κοινοβούλιο πρέπει να εφαρμοστούν το κοινοβούλιο μας δεν ε, έλαβε ποτέ θέση στα εσωτερικά ε, πολιτικά πράγματα της Μάλτα. Εμείς θέλουμε να δούμε ποιος δολοφόνησε τη Δάφνη. Προχωρούμε τώρα. Παρακαλώ, σεβαστείτε την κανονική ε, λειτουργία του Κοινοβουλίου. Μην ζητάτε διαδικαστικά. Έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες. Και άλλο διαδικαστικό τώρα. This is going to be the last point of order. Το τελευταίο όμως, γιατί έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες. Παρακαλώ δεχτείτε την κανονική διαδικασία. Σύντομα. Ναι, μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομη, κυρία Νετφέλτ, και μιλώ ως πρόεδρος ε, της ομάδας που παρακολουθεί το κράτος ε, δικαίου. Συνεδριάσαμε σήμερα το πρωί. Προγραμματίζουμε επίσκεψη στη Μάλτα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία πολιτική παρέμβαση, ούτε θέλουμε να πάρουμε το μέρος κανενός, ούτε να ανακατευθούμε στις έρευνες της αστυνομίας, ούτε στη δικαιοσύνη, αλλά να βεβαιωθούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να κρατάει την πίεση εκεί ε, ε για να καταλάβουμε και να βρούμε τι έγινε τέλος πάντων κάποια στιγμή. Και τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Πρώτο σημείο, κοινό ψήφισμα για την κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία. Τροπολογία 1, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε δυνάτες στις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενο. Κατάσταση στην Κούβα η περίπτωση του Χωζέ Ντανιέλ Φερέρ. Πρώτη παράγραφο, αρχικό κείμενο, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα το ψήφισμα συνολικά έρχεται ψηφοφορία ονομαστική κλίση. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενο, IT, κοινό ψηφίσμα πέντε πολιτικών ομάδων. Διανάταση χειρός ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο. Έκθεση Λάγκε. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενο. Ψήφισμα που συνοδεύει την προηγούμενη έκθεση. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρία Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφορία. Ονομαστική κλίση. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα συνολικά διανάταση ισχυρό υπέρ. Με συγχωρείτε ονομαστική κλίση, δικό μου το λάθο. Πιέστε τα κουμπιά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Το ψήφισμα εγκρίνεται. Επόμενο, κατάσταση στην Βολιβία. Κοινό ψήφισμα τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Τροπολογία 1, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2, ονομαστική κλίση, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Διανάταση ισχυρός. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Διανάταση ισχυρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχο. Παρακαλώ ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα το ψήφισμα συνολικά όπως τροποποιήθηκε ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. What is Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα, κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τροπολογία 10. Διαδικαστικό, παρακαλώ. Microphone, please. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια υπενθύμηση για τον εσωτερικό κανονισμό. 132 εδάφιο 2 του εσωτερικού κανονισμού προβλέπει ότι επειδή τη Δευτέρα το βράδυ είχαμε συζήτηση για την κατάσταση εκτακτή ανάγκη του κλίματο και του περιβάλλοντο, είχαμε την αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε στον τίτλο τον όρο «κατεπήγων», ενώ υπάρχουν ανατροπολογίες που προτείνουν να χρησιμοποιήσουμε τον όρο απλώς επίγων. Emergency σε αντίθεση με το urgency. Εδώ λοιπόν οι τροπολογίες αυτές που προτείνουν την αλλαγή στον τίτλο πρέπει να θεωρηθούν μη παραδεκτές. So the title of the... Ο τίτλος της συζήτησης δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από τον τίτλο του ψηφίσματος. Μάλλον μπορεί να είναι διαφορετικός από τον τίτλο του ψηφίσματος. Οπότε τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχο. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Έλεγχο για τη 10. Άρχεται. What is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Amendment 7. 7. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τοπολογία 11, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ω, με συγχωρείτε, δυνάταση ισχυρό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία. Αρχικό κείμενο, λοιπόν. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση. Ωραία. Έλεγχο. Έλεγχο για το 9. Τροπολογία 9. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ωραία. Αρχικό κείμενο λοιπόν σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Διανάταση χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, διονομαστική ε, κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. 15. 15. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική κλίση. Λειτουργούν τώρα. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική κλίση. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία πρώτη. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα αρχικό κείμενο. Αιτιολογική αναφορά 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το ψήφισμα ως σύνολο. Διανομαστικής κλίσης. Άρχεται η ψηφορία. Ονομαστική κλίση. Ωραία, ηλεκτρονικά. Πέρας. Το ψήφισμα εγκρίθηκε. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρος. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Και τώρα έχουμε την πρόταση ψηφίσματο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η κυρία Βυσνιεύσκα, έχει ζητήσει το λόγο. Όχι, η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με το 139 θα ήθελα να πω ένα διαδικαστικό γιατί πρόκειται περί τροπολογίας που από κοινού κατεβάσαμε με άλλες πολιτικές ομάδες αλλά με αίσθηση ευθύνη. Πρόκειται να απόσχουμε. Πρόκειται για την τροπολογία 11 που αφορά για την επίγουσα κατάσταση σχετικά με το κλίμα. Γιατί υπάρχουν κάποιες πολιτικές ομάδες που θέλουν να θάψουν το κείμενο λόγω αυτής της τροπολογίας. Αφού μιλούμε για επίκουσα κατάσταση δεν είναι δυνατόν να διαγενερεύσουμε το κείμενο για το COP25. Θα πρέπει όλοι μαζί και το ΕΛΚ να εμφανιστούμε ενωμένοι με το ψήφισμα για το COP25. Κύριε Βεσίνιαυσκα, έχετε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αποσύρω την υποστήριξή μου αλλά και την υποστήριξη του ECR για το ψήφισμα αυτό που αφορά το COP, την COP μάλλον 25. Δεν θέλουμε να γίνει η συνάντηση πιο νωρίς. Έχουμε το κατόφλι αυτό το καινούριο του 55%. Πέραν αυτού, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου θέλει να δώσει το πράσινο φως στην πυρηνική ενέργεια. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ κακό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό δεν βρίσκει σύμφωνα τα μέλη. Ψηφίζουμε, λέει η Πρόεδρος. Επομένως, πρόκειται για τη διάσκεψη την κλιματική αλλαγή. COP25. Ψηφίζουμε με Ονομαστική κλίση. Πέρασε ψηφορίες. It's rejected. Και απορρίπτωται. Τροπολογία 51. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρασε. It's rejected. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στο αρχικό κείμενο. Δεύτερο τμήμα. Με ανάταση χειρός υπέρ το πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση ψηφίζουμε πέρασε εγκρίνεται 52 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε πέρασε Εγκρίνεται. Παραγραφός 9 του αρχικού κείμενου εις τρία τμήματα. Το πρώτο ονομαστε κύκλιζε. Ψηφίζουμε. Πέρασε. It's adopted. Second part by showing... Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ανάταση χειρός υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14 του αρχικού σε δύο τμήματα, το πρώτο ονομαστική. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, ανάταση χειρός υπέρ, κατά, α, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 20 αρχικό κείμενο, το δύο τμήματα, το πρώτο υπέρ, κατά, α, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται ηλεκτρονικός έλεγχος για το 43 ψηφίζουμε πέρασε απορρίπτωται το αρχικό κείμενο τώρα. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα με ανάταση χειρός υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 44 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 45. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα. 53. Σε δύο τμήματα το πρώτο. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Πέρασε. It's rejected. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ανάδας χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία υπερθμών 1. Ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτονται. Τροπολογία 19. Ονομαστική. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Α, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, σε δύο τμήματα, το πρώτο. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ. Ανάταση χειρός. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 ονομαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο. Ονομαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ να τα συγχυρός. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. What is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 26. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ανάταση χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 28 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Ανάταση χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στο αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Check. Check, check. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου. Πέρας. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο. Ονομαστική κλίση. Παράγραφος 33. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Υπέρ. Ανάταση χειρός. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 58. Ονομαστική κλίση. Υπέρ. Πέρας. Και απορρίπτεται. 59. Ανάταση χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Με ανάταση χειρός. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 μονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60, ανάταση χειρός, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για το 60. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εξήντα ένα. Ανάταση χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Με ανάταση χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Το 37. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα, το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Το πρώτο με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με να τα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Σε δύο τμήματα το πρώτο. Ονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Πέρασε. Ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Κάποιον οι τροπολογίε 10 και 63 και πάμε στην τροπολογία 4 με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε. «52, παράγραφος 4, ονομαστική κλίση. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 64 με τα συγχυρώσει. υπέρ κατά Αποχέ. απορρίπτονται Ηλεκτρονικό έλεγχο το 64 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτονται 65 υπέρ Ανάταση χειρός. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Είπαμε επόμενη καταπίπτει και πάμε τώρα στην τροπολογία 23. Υπέρ. Ανάταση χειρός. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 47, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Και πάμε στην παράγραφο 54, το αρχικό κείμενο. Ανάτας χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το Τοπολογία 38. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. We go to 58 αρχικό κείμενο. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ. Ανάταση χειρός. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Για το 58, πρώτο τμήμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Ανάταση γύρω. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 48, με ονομαστική κλίση. Θέλετε να γίνει έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 58, δικαιούστε να το ζητήσετε, 58, δεύτερο παράγραφος, δεύτερο τμήμα μάλλον. Ε, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. 58, δεύτερο τμήμα. Γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος, πέρας. Απολύπτωτο. Τροπολογία 48. μας κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 66 υπέρ, για να χειρός. Κατά. Άποχες. Θα ήθελα να κάνω ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε. Πέρας. απολύτως. Αρχικό κείμενο. Σε τρία τμήματα. Το πρώτο. Με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. είπε. Ανάταση χειρός. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 64, το αρχικό κείμενο, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24, υπέρ. Κατά. Αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για το 24. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 σε δύο τμήματα. Το πρώτο με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 67. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 12 και 26 σε δύο τμήματα. Το πρώτο, ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Με ανάταση χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στο αρχικό κείμενο. Υπέρ. Με ανάταση χειρός κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 13 και 27 με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στο αρχικό κείμενο. ποιοι είναι υπέρ με ένα Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία, ε, τροπολογίες 14 και 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Οι 15 και 29. Υπέρ, υπέρ, υπέρ, υπέρ. Συγγνώμη. Ξανά, ξανά. Οι 15 και 29. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Οι τροπολογίες 16 και 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Η τροπολογία 31D με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 6 με ονομαστική κλίση αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 9. Το αυτόν. Άρχιτη ψηφοφορία. Ονομαστικά πάντα. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 32. Ονομαστικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα το αρχικό κείμενο καταπίπτει, οπότε και θα πάμε στην παράγραφο 69, τροπολογία 34. Δυνατά χειρός υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες. Έλεγχος. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 34. Συγγνώμη, 69 της παραγράφου, το αρχικό κείμενο. Πέρας. Κρίνεται. Οι τροπολογίες 18 και 35 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον, υπέρ. Οπ. Θέλετε παλήθευση. Uh, point of order. Διαδικαστικό, κύριε Ταραμπελά. Τι θέλετε. Έχετε το λόγο. Δεν θέλω να παρατείνω τις ψηφοφορίες. Μια πρόταση να κάνω ε, για τους επισκέπτες μας, για τη βολή τους. Όταν έρχονται ε, οι επισκέπτες, όπου και να κάθονται, τα καταλαβαίνουν όλα να έχουμε συζητήσεις. Στις ψηφοφορίες όμως όσοι κάθονται απέναντί σας καταλαβαίνουν τι γίνεται και βλέπουν και ε, τους πίνακες προτείνω να βάλουμε πίνακα και απέναντι για να καταλαβαίνουν όσα συμβαίνουν όσοι κάθονται πίσω σας. Thank you very much for your We'll... Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Ε, θα το εξετάσουμε. 18 και 35. Ε, είμαστε σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο Τσεκ. Καλά. Επαληθεύουμε λοιπόν ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα. Στι τροπολογίες 15, 18 συγγνώμη, και 35. Πέρα. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τώρα απορρίπτεται. Τροπολογία 68. Τι τσεκ. Τσεκ. Ωραία. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Αρχίζει ψηφοφορία. Τροπολογίες 18 και 35. Τμήμα δεύτερο. Πέρασε. Απερίφθη. Η τροπολογία 68 σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, διανατάσεως της χειρός υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Στην τροπολογία 69 είμαστε τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 36 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Στην 36 παρακαλώ αρχίζει ψηφοφορία. What is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 50 καταπίπτει. Και ερχόμαστε στην τροπολογία 70. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Ε, ε, επαλήθευση. Είναι μικρές οι διαφορές. Πέρας. Ε, όχι και τόσο. <laughs> Κρίνεται. Καλώς. Η τροπολογία 70. Ψήφι υπέρ. 70. 70 we did. I'm sorry. Α, όχι, την κάναμε. Ωραία. 7D. 7D. Ζητώ συγγνώμη. Ε, φταίει ο δαίμον του τυπογραφείου. Δεν είναι 0, είναι D και το είδα για 0. 7D ε, με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Το βρήκαμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 8D. ο ισχυρό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε στην παράγραφο 77 το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Καλά. Στην παράγραφο 77 το δεύτερο τμήμα ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία και τελειώνει. Εγκρίνεται. Παράγραφος 78. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο είναι με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 80. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο διανατάσσεω χειρό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 82 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο, υπέρ, ε, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα ονομαστικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 83 του αρχικού κειμένου υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Παράγραφος 90 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Παράγραφος 91 το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στην τροπολογία 71. Ψηφί υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 72 με νομαστική κλίση αρχίζει τώρα. What is closed? Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 115, το αρχικό κείμενο ψηφίπερ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο με ονομαστική κλίση αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 118 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η, η τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές Ας το επαληθεύσουμε αυτό σας παρακαλώ. Τροπολογία 39. Πέρασε. Εγκρίνεται. Μητροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ιδεολογική σκέψη γιώτα. Υπέρ. Όχι ένα, όπως είχε πει η Πρόεδρος. Ακόμα δεν τα έχω μάθει. Άι, γιώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Η αιτιολογική σκέψη K. Λατινικό. Με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη L. Η τροπολογία 42 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ. Τσεκ. 42. Τροπολογία, τμήμα πρώτον, Ελεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ψηφίζουμε ονομαστικά το, την πρόταση ψηφίσματος της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ECR. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στο ψήφισμα του ECR. Πέρασα. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 4, ονομαστικά. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7 του αρχικού κειμένου, ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3. Ονομαστικά. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 2. Και πάλι ονομαστικά. Vote is open. Vote is now closed. Πέρασε. Απορρίπτεται. Και τώρα η αιτιολογική σκέψη L του αρχικού κειμένου ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Now we go to the next... Προχωρούμε. Επόμενο θέμα προς ψήφιση. Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών. Κοινή πρόταση ψηφίσματος πέντε πολιτικών ομάδων. Ψηφίζουμε το σύνολο με ονομαστική κλίση. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα. On our agenda. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η διένεξη της διαφορά της Airbus. Τέσσερις πολιτικές ομάδες έχουν καταθέσει ένα κοινό ψήφισμα. Η τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η παράγραφος 7, το σχικό κείμενο σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ, κατά, απόχες εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 4, υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 11 ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 3 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 υπέ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 10 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και τώρα το σύνολο του ψηφίσματος, διανατάσσεως χειρός υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. We go Προχωρούμε. Ε, στο επόμενο θέμα, η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιωτικό όργανο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Η τροπολογία 2, ονομαστικά. Είναι ένα ψήφισμα της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου. τα. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 1, διανατάσεις της χειρός είπε κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και το σύνολο του ψηφίσματος, ονομαστικά παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα, τελευταίο θέμα ε, είναι ε, το ψήφισμα για τις ενεξέλεξη διαπραγματεύσεις ε, με την ΑΚΕ. Παράγραφος 17, πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές έλεγχος στην τροπολογία παριθμών 1. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Θέλετε έλεγχο επαλήθευση της πρώτης λοιπόν, του πρώτου τμήματος. Ε, τροπολογία 2, τμήμα 1, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. Okay, now we go to the second. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει, οπότε η τροπολογία 5 υπέρ. Όχι. Yes, and now we go to the amendment 5, yes. Ναι, πρέπει να ψηφίσουμε την 5, σωστά, αφού έχει καταψηφιστεί η προηγούμενη. The second, because the first part is rejected, so the second part falls. Καταψηφίστηκε το πρώτο τμήμα, κατέπεσε το δεύτερο, άρα ψηφίζουμε την τροπολογία 5 τώρα. Ο ψήφι Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Και τώρα το αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση, η οποία αρχίζει και τελειώνει. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ε, διανατάσσεως ισχυρό τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται και η τροπολογία 4 υπέρ, κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ και για την υποστήριξή σας. We have minutes. We have minutes and... Δύο λεπτά διάλειμμα για να συνεχίσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. Παρακαλώ, αποχωρήστε γοργά.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 before you start calling the names that you say Let's continue because we have very little time left and a lot of people would like to take Συνάδελφοι, παρακαλούμε να καθίσετε για να ξεκινήσουμε, γιατί είναι πολύ που έχουν ζητήσει το λόγο για τι επεξηγήσει ψήφων. Παρακαλώ, σε περίπτωση που δεν θέλετε να ε, συμμετάσχετε, να αποχωρήσετε. Παρακαλώ, αν θέλετε τα πηγαδάκια έξω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, θέλετε να τα πείτε τα ιδιαίτερά σας εκτός αίθουσας και τις φωτογραφίες επίσης εκτός να προχωρήσουμε σε επεξηγήσεις ψήφων από χθες, αυτές που δεν μπόρεσαν να καλύψουν χθες και μετά θα περάσουμε στις επεξηγήσεις για τη σημερινή το σημερινό γύρο ψηφοφοριών. Να σας πω ότι έχουμε πολλές προφορι πολλά αιτήματα για προφορική επεξήγηση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε γοργοί, γιατί στις δύο πρέπει να αποχωρήσουμε από την ε, αίθουσα της Ολομέλεια. Να παραμείνετε στο μονόλεπτο, παρακαλώ. Ε, ό,τι απομείνει μπορεί να υποβληθεί γραπτός. Πρώτον, εκλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επεξήγηση ψήφων, χουκ από την ομάδα Ρινιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το γεγονό ότι εξελέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαίνει ότι η λογοδοσία τη στο Κοινοβούλιο εξακολουθεί και αυτό είναι ζωτική σημασία. Οι υποψήφοι που προτάθηκαν από τι κυβερνήσει των όλων των κρατών μελών ε, πέρασαν από ακρόαση και εγκρίθηκαν τελικά. Πρέπει να ξεκινήσει να δουλεύει η Επιτροπή. Είναι πολλοί ο κόσμο που περιμένει τη βοήθειά μα. Ε, κόσμο που ε, απειλείται από του κινδύνου των κλιματικών αλλαγών, από τι αβεβαιότητε τη μεταβαλλόμενη οικονομία. Κόσμο που αισθάνεται αδύναμο στην καθημερινότητά του να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Η δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να δώσει σε όλου τα όπλα για να μπορούν να αντικρίσουν το μέλλον με ελπίδα και όχι πλέον με φόβο. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρήσει στο ε, σφάλμα του Brexit και χαθεί φωνή μα από την Ευρώπη, οι αποφάσει που λαμβάνονται εδώ και πάλι θα ταράσουν το μέλλον και θα χαράζουν το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Ω Βρετανό βουλευτή, λοιπόν, ήθελε να εκλεγεί το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχα την ελπίδα ότι θα ε, ανακοπεί η πορεία προ τον Brexit. Προ όφελο όλων των Ευρωπαίων Ευχαριστούμε κύριε Ζάχραντιλ από την ομάδα συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαδευτεί από την ιστερία για το κλίμα που είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα και η οποία έχει ρίξει βαρύ ίσκιο στην όλη διαδικασία εκλογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών είναι σίγουρα ε, ε, έτσι όπως προτείνεται σήμερα ανέφικτη και είναι και επικίνδυνη για τις εθνικές οικονομίες μας. Επηρεάζει το ενεργειακό μείγμα, τις δομές, την απασχόληση και γι' αυτό ακριβώς δεν μπόρεσα να υποστηρίξω την εκλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε κυρία Βρετσόνοβα από τους Ιδρυτικούς και Μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε με την ψήφο μου ε, δεν ε, ψήφισα υπέρ της, εκλογή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως προτείνεται, διότι το πρόγραμμα εργασιών της είναι τοπικό. Απειλείται ανταγωνιστικότητα της επίρου μας, ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ωραίο να συμπεριλαμβάνουμε το στόχο των ακτιβιστών, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν στην πραγματικότητα. Εάν του πετυχάναμε, θα καταστρέφαμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία, θα αυξάναμε τι τιμέ τη ενέργεια και θα δημιουργούσαμε δυσφορία στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών οι αγορέ θα καταστραφούν και τα μερίδια αγορά των ευρωπαϊκών εταιριών θα τα πάρουν οι κινέζικε και αμερικάνικε. Χωρί κανέναν έλεγχο. Η πράσινη αυτή επανάσταση είναι κάτι το πανάκριβο που θα πρέπει να το πληρώσουν, να πληρώσουν τελεπιτεροί οι δικοί μα φορολογούμενοι. Ε, είμαστε οι μόνοι που θέλουμε να πάρουμε τέτοια μέτρα. Ευχαριστούμε κύριο Ρόρι. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ήταν μακράν το τέλειο η διαδικασία που έγινε τους τελευταίους ε, μήνε όμω. ήταν πάρα πολύ σημαντικό διότι μα έδωσε την ευκαιρία να αλλάξουμε την γνώμη μα σε σχέση με αυτό που ψηφίσαμε τον Ιούλιο όσον αφορά τον ε, ορισμό τη Πρόεδρου Φοντερ και κατόπιν είχαμε κάμποσε εβδομάδε για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τι λεπτομέρειε του προγράμματο εργασιών και να μπορέσουμε να το αναλύσουμε και να υποβάλουμε τι ενστάσει μα στην Επιτροπή που χθε την ε, ψηφίσαμε και πρόκειται για ψήφο επιβεβαίωση σε σχέση με ό,τι ψηφίσαμε τον Ιούλιο. Αλλά εγώ σας προτείνω ότι αυτό το, να δίνεται δηλαδή ευκαιρία του να σκεφτεί κανεί τι αποφάσει προηγουμένω είναι κάτι το σημαντικό και αυτό θα πρέπει να αφορά και άλλα ζητήματα και αλλού. Σε ευχαριστούμε κύριο Σκανάν από το ECR. Ευχαριστώ ε, κύριε Αντιπρόεδρε. Είναι πάρα πολύ φροντισμένα είναι όλα αυτά ε, και σε λίγο αυτό δεν θα μας αφορά εμάς. Ναι, αλλιώς αν θα μπορούσαμε πολλά να πούμε επί της ε, ουσίας. αλλά τέλος πάντων πολλά θα μπορούσαμε να πούμε όσον αφορά αυτή τη διαδικασία του ορισμού των επιτρόπων, αυτού της συγκέντρωσης νομοθετικής εξουσία, ε, νομοθετικής εξουσίας σε αυτούς οι οποίοι είναι μακράν των εκλογών, και οι οποίοι είναι θωρακισμένοι από την κοινή γνώμη. Αλλά τέλο πάντων αυτό δεν θα είναι το πρόβλημα μα λίγο. Οπότε ευχόμαστε καλή επιτυχία και περιμένουμε πώ και πώ να γίνουμε αντί για δύσκολοι συνεργάτε να είμαστε καλοί γείτονε και καλή τύχη. Κύριε Λεμπρετών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα κατά τη άνοιξη καθηγόντων και στον γιατί νομίζω ότι η κατάσταση θα γίνει χειρότερο όσον αφορά την ε, Γαλλία σε τρει βασικού τομεί. Πρώτα, πρώτα είναι η υπέρ τη μετανάστευση ε, στην Ευρώπη, όμω πρέπει να κάτι άλλο, να υπάρξει καταπολέμηση κατά αυτή τη πλημμυρίδα των μεταναστών. Επίση θέλει να μα εξαναγκάσει σε ολοκλήρωση, Εμεί όμω, στη, πάρα πολύ από εμά, ο εθνικό συναγερμό ε, ζήτησε εθνική κυριαρχία. Επίσης θέλει να συνεχίσει αυτήν την τρελή πολιτική της παγκοσμιοποίηση του για των ελευθέρων συναλλαγών και αυτό θα χτυπήσει την Γεωργία και για αυτούς του τρεις λόγους εγώ είμαι κάθετα εναντίον της Επιτροπής Φόντερ Λάιν και αυτό θα το υποστήριξω σε όλη μου την θητή. Ευχαριστούμε κυρία Φόξ. Μία γεγραμμένη. Εγώ ψήφισα κατά Κατά, κατά. Κατά της Νέας Επιτροπής. Διότι να λέμε ότι εξελέγει είναι λάθος. Δεν είναι υπόλογοι στους ε, ψηφοφόρους. Από καμία χώρα υπονομεύει την εθνική κυριαρχία. Πρόκειται για μια προσβολή προς κάθε υποψήφιο. Λένε ότι είμαστε ακροδεξιοί, ότι είμαστε ξενόφοβοι. Ε, όλα αυτά είναι συκοφαντίες. Αυτό είναι ένας φερετζές νομιμοποίησης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ελληνική σημαίνει σεβασμό των ψηφοφόρων παντού στην Ευρώπη. Παρακαλώ οι συνάδελφοι δημοκράτες ε, ευρωβουλευτές να μην κάνουν ότι εδώ είναι δημοκρατικός χώρος γιατί δεν έχουν καμία σχέση οι με αυτά. Χρειάζεται να είναι κανείς ε, υπόλογος ψηφόρος του. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να το πράξουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα το Κοινοβούλιο έχει ε, ακολουθήσει πλήρως, ε, τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, διότι απομακρύνθηκαν οι υποψήφοι οι οποίοι λόγω σύγκρουσης συμφερόντων είχαν ε, απορριφθεί και βρέθηκαν καινούργοι. Ε, γι' αυτό η νέα επιτροπή μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη. Και το πρόγραμμα εργασιών τη είναι αξιόπιστο και για άλλου λόγου. Διότι αναζητά αποκρίσει ε, στι. Ε, στι κρίσει που έχει αποφύγει τώρα το Συμβούλιο, τι κλιματικέ αλλαγές και άλλα μέτρα για την ψηφιακή αγορά, κοινωνική δικαιοσύνη, όλα αυτά είναι λόγοι, ε, των οποίων ψήφισε υπέρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θέλουμε κι άλλο μισό χρόνο καθυστέρηση, ούτε να προκαλέσουμε χάος και ματαιώσεις. Ε, έχουμε ήδη χάσει πολύ χρόνο από τη θητεία μας, γι' αυτό ψήφισε υπέρ της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε κύριος Ολέκας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστήριξα την ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ψήφο μου, διότι υποστηρίζω την Πράσινη Συμφωνία. Χρειαζόμαστε το Green Deal για να επιβιώσουμε. Το χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Επίσης, υποστηρίζω την ψηφιοποίηση, την καινοτομία και θέλω να υποστηριχθούν οι περιφέρειές μας μέσω της γεωργίας και της κτηνοτροφία. Θέλουμε ίσες αμοιβέ για τους γεωργού σε όλε τις χώρες, ιδίω στα κράτη της Βαλτική η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και για το όφελο των ε, ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και για να οδηγήσουμε και τι γειτονικέ μα χώρε, τι χώρε τη Αφρικανική Υπήρου. Χέρι-χέρι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα και να τηρήσουμε τι υποσχέσει που δώσαμε στου Ευρωπαίου ψηφοφόρου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, αλλά λόγω τη προφορική επεξήγηση δεν ε, προβλέπει ο κανονισμό ε, διαδικασία γαλάζια κάρτα. Με συγχωρείτε, αλλά είχα ζητήσει το λόγο, αλλά δεν βλέπω το όνομά μου στην οθόνη. Δεν ήθελα να, να διακόψω κανέναν, ούτε να ε, ζητήσω το λόγο με γαλάζια κάρτα. Μα είχατε υποβάλει έτοιμα για να πάρετε το λόγο. Ναι, κατάλαβα μάλιστα ότι είχε επιβεβαιωθεί, αλλά δεν με βλέπω στην οθόνη. Εντάξει, αν προλάβουμε θα σας δώσουμε το χρόνο. Ο κύριος Πάτεν από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ. Εγώ καταψήφισα την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πιστεύω ότι ο διορισμός της το ε, δείχνει ε, και επιβεβαιώνει ότι είναι ρατσιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θεσμικά. Το 10% των Ευρωπαίων πολιτών είναι χρωμή και δεν είχαμε δει ποτέ μαύρο επίτροπο, ε, ούτε σε ηγετικέ θέσει στην διοίκηση. Οπότε δεν έχει εκφραστεί εδώ η διαφορετικότητα. Δεν είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία εδώ. Είμαστε apartheid. Την ημέρα Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για τους λευκούς. Το βράδυ ανοίγουμε τις πόρτες στους μαύρους για να σφουγγαρίζουν ε, τα πατώματα και να καθαρίζουν τις τουαλέτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να έχει ε, έχρωμους μαύρους. Επέμενε για γυναίκες η κυρία Φόντερ Λάιν. θα μπορούσε να έχει επιμείνει και για τους μαύρους και να προσλαμβάνονται περισσότεροι μαύροι. Ο πρόεδρος εχθές μίλησε για αλλαγή του προσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βέβαια πάντα στο βαθμό που παραμένουν λευκά τα πρόσωπα αυτά. Εγώ δεν ε, ψηφίζω αυτούς τους λευκούς δουλεμπόρους. Ε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπάντινγκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ως Βρετανή Ευρωβουλευτής είμαι υπερήφανη που ε, είμαι από μια κυρίαρχη χώρα που ε, συνεργάζεται με τους εταίρους μας στην Ευρώπη για ε, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Έχει εξαντλήσει στην Ευρώπη μια σειρά από δήμους και περιφέρειες την έκτακτη ανάγκη για το κλίμα. Σήμερα όμως στην Ήπειρο δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση άμεση για να αναστρέψουμε τις ζημίες που έχουν προκληθεί στον πλανήτη πριν τελειώσει ο χρόνος, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Θα πρέπει όλοι να μειώσουμε το αποτύπωμα αντιοξιδίου του άνθρακα από την τροφή μας, από την τεχνολογία μας, από τους ωκεανούς, από το εμπόριο και τις εισαγωγές μας. Μαζί θα πρέπει να εργαστούμε και θα το κάνουμε για να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παγκοσμίως. Η αλλαγή αρχίζει από εδώ. Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι προφορικές ε, επεξηγήσεις ψήφου για τον προϋπολογισμό του 2020. Το λόγο έχει ο κύριος Άχραντήλ από την ομάδα ECR. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πριν από λίγο επέκρινα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κλιματική της πολιτική και τώρα για αλλαγή ε, θα την επενέσω για τα σχέδια που έχει ε, σχετικά με την επόμενη περίοδο και τον προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά ε, τις μεταφορές πιστώσεων και τις μεταβιβάσεις. Φεύγουμε από τις άμεσες επιδοτήσεις και τις άμεσες ενισχύσεις της πολιτικής συνοχής και της γεωργίας και υποστηρίζουμε την έρευνα ε, και τους επιστήμονες. Δυστυχώς αυτό ακόμα δεν αντανακλάται στο ε, Κοινοβούλιο γιατί εμεί συνεχίζουμε το χαβά μα. Θα ήταν όμω καλή ιδέα να στείλουμε ένα μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα επιμείνουμε σε αυτέ τι δεσμεύσει που ανέλαβε ε, εχθέ η κυρία Φόντερ στην παρθενική τη ομιλία. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την έκθεση αυτή γιατί δεν είμαι σύμφωνος με τους προσανατολισμούς του προπολογισμού. Βρετσιόνοβα, κυρία Πρόεδρε, Ούτε εγώ μπορούσα να ψηφίσω υπέρ αυτού του προπολογισμού χθε, γιατί έχουν ανέβει τα έξοδα, οι δαπάνε και που γίνονται σε κάποιου τομεί που είναι τελείω άσχετε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βελτιώνουν την ανταγωνιστικά τη Ένωση ή των κρατών μελών. Πρόκειται για διασπάθηση του χρήματο του φορολογουμένου. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να υποστηρίξει κανεί θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικές κάποιες επιδοτήσεις σε κάποιους τομείς, μα αυτές είναι όμως επιζήμιες και ενώ διάφορες ε, εταιρείε που δεν βγάζει νόημα αυτή η πολιτική, δεν συμφωνώ. Κύριο Χάναν, έχει δει στο λόγο, αλλά δεν είναι εδώ. Οπότε πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η Βολιβία. Κύριε Πόσπη λέγεται τον λόγο. Ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά ψήφισα υπέρ αυτού του κειμένο στην ε, τελευταία θητεία. Συζητήσαμε πολλές φορές για τη Βολιβία και μιλήσαμε για την πολιτική Μόραλες και είχαμε διατυπώσει ανησυχία και υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσον ε, είναι δίκαιες ε, οι εκλογές. Τελικά αυτός ο δικτάτορας δραπέτευσε, έφυγε από τη χώρα και στη Βολιβία η Βουλή ετοιμάζει νέες ελεύθερες εκλογές. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να μας χαροποιήσει και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσέξουμε αυτές οι εκλογές να γίνουν χωρίς νοθείες. Και έτσι να βελτιθεί η κατάσταση στη χώρα. Ευχαριστώ λέει Και τώρα το επόμενο θέμα είναι κλίμα και περιβάλλον. Και έλεγχε. Ρινιού. Ευχαριστώ. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η ζήτηση των τελευταίων εβδομάδων και το θέμα είναι σοβαρό. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια μας. Τα επιστημονικά δεδομένα είναι γνωστά. Θερμαίνεται ο πλανήτης. Έχουμε όλες αυτές τις ε, εκπομπές από τα καύσιμα και γι' αυτό και χρειάστηκε επιγόντως κάτι να κάνουμε για αυτό το ψήφισμα. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις νέες γενιές, αυτές τις χιλιάδες των ανθρώπων που την Ιρλανδία κάθε Παρασκευή κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα, γιατί πρέπει να προστατεύσουν περισσότερο οι πολιτικοί και οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Άρα τώρα θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι το πράγμα επήγει και άρα κάτι να κάνουμε κάτι να κάνουμε επιγόντω από πλευράς χάραξη πολιτικών που θα έχουν άμεσα αποτελέσματα να σώσουμε τη γη, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τους ωκεανούς. Έχει παραγίνει το δεν είναι θέμα αν είναι επίγον ή κατεπίγον. Είναι αυτό που είναι, που φαίνεται τι είναι. Άρα χρειάζονται πολιτικές που θα λύσουν το πρόβλημα. Πάλμερ, σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Εγώ δεν πιστεύω ότι το ψήφισμα που πέρασε σήμερα για την κλιματική κατεπίγουσα έκτακτη ανάγκη ε, θα μπορούσε να είχε εγκριθεί αν δεν υπήρχε η καμπάνια και η πίεση όλων αυτών των χιλιάδων νέων παντού στον κόσμο που διαδηλώνουν, που ε, φεύγουν από τα σχολεία τους, από τα γυμνάσια και από τα λύκια για να διαδηλώσουν. Και την περασμένη εβδομάδα με χαρά ήμουν και εγώ στη διαδήλωση. Αυτό που τους νοιάζει δεν είναι εμείς να ε, εγκρίνουμε ψηφίσματα, δεν θέλουν λόγια. Έργα θέλουν, αποφασιστική δράση και τίποτα άλλο. Και αυτό τώρα θα πρέπει εμείς να τους δώσουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα ε, κράτη και οι κυβερνήσεις μας αλλά και εμείς ως Κοινοβούλιο. Τώρα έχει έρθει η ώρα για έργα. Γιατί τι μας λένε αυτοί οι νέοι. Και η Γκρέτα Τούμπερκ όταν μίλησε εδώ στο Κοινοβούλιο πριν από λίγους μήνες. Δεν αρκούν τα λόγια. Δράση θέλουν οι νέοι μας και έχουν δίκιο που απαιτούν ε, δράση από εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φόξ, μία εγγεγραμμένη. Εγώ καταψήφισα αυτό το ψήφισμα ε, για την κατεπήγουσα έκτακτη ανάγκη, γιατί ε, Αυτά είναι ε, κινδυνολογίες για να τρομάξει ο κόσμος ε, ότι θα καταρρεύσει ο πολιτισμός και τα λοιπά. Και ε, όλα αυτά τα προωθεί η ΜΚΟ Extinction Rebellion. Είναι αντιεπιστημονικά και οι τελευταίες μέρες έδειξαν τη συζήτηση. Καταψηφίσαμε λοιπόν αυτές τις τροπολογίες που έλεγε ότι θα πρέπει να δεσμευτούμε, να ξαναφέρουμε τη συζήτηση σε λογικά πλαίσια. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστερία είναι προπαγάνδα, δεν είναι επιστήμη πια. Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία από την IPCC ή οποιονδήποτε άλλον για την ε, εξαφάνιση και τον αφανισμό της ανθρωπότητας. Δεν θα πρέπει να λέμε ότι είναι ανθρωπογενείς οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και όλα αυτά που ζούμε. Ε, τυχαία τις τελευταίες μέρες. Η Επιτροπή IPCC έχει πει ότι ε, αυτά είναι κοινωνικο-οικονομικά αίτια θα έχουμε λιτότητα φεύγοντας από τον άνθρακα, τεράστιες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και όλα αυτά τα κάνουν για να τρομακρατήσουν τον κόσμο. Ευχαριστώ παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης. Ο κύριος Ρόλαντ ε, μου φαίνεται ότι έφυγε. Α, όχι. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε ο συνάδελφο και εγώ απορρίπτω το ψήφισμα για την COP25. Ε, Μπορεί να μην είμαι καθηγητής, δεν χρειάζεται ε, για να καταλάβω οικονομικά και για την επιστήμη. Ε, τα δεδομένα για τι αποκαλυπτικέ αυτέ προοπτικέ με την κατάσταση Έκτακτη ανάγκη των περιβάλλων, ούτε αυτά τα πιστεύω γιατί ουσιαστικά πρόκειται για παραδείγματα ε, α, ε, πλήρους άγνοιας ε, και προσπάθειας εκφοβισμού. Πρέπει ε, να μελετήσουμε τη μελέτη επιπτώσεων για τις κλιματικές αλλαγές. Για το καθαρό μηδέν πραγματικά φαίνεται να είναι ψίχουλα, ψίχουλα επιπτώσεις του Brexit ε, σε σχέση με αυτό πρέπει να γίνει για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί για το ότι πρόκειται για μια τεράστια μηχανική, ε, ένα μηχανικό εγχείρημα που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο. Εκτός από περιόδους πολέμου δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ένα τρισεκατομμύριο αγγλικές λίρες, 2% του ΑΕΠ το χρόνο είναι αυτά που απαιτούνται με αυτή την τρελή πολιτική που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ κύριε Σομαρζέ, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα 28 Νοεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίες κατάκταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και το περιβάλλον. Είναι συμβολική αυτή η στιγμή και ιστορική. Είμαι υπερήφανος ε, που συνεισέφερα σε αυτό με τη δική μου ψήφο. Η Ευρώπη μετά τη βιομηχανική επανάσταση ουσιαστικά συνεισέφερε στην ε, καταστροφή του κλίματος. Έχουμε λοιπόν χρέος και καθήκον απέναντι στους λαούς του κόσμου στα διάφορα είδη της παπανίδας, της χλωρίδας και ιδίω όμως απέναντι στους νέους μας που μας ζητούν να δράσουμε σήμερα. Ναι, πρέπει να δράσουμε σήμερα για να μπορεί κανείς να ζει στον πλανήτη Γη και στο μέλλον. Τόσο άνθρωπος όσο και όλα τα άλλα είδη που απειλούνται με αφανισμό. Είναι κάτι πρωτόγνωρο όλο αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε άλλο. Πρέπει να δράσουμε. Ευχαριστώ κυρία Σόντροβα. Από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να μιλήσω ακριβώς για το θέμα μας της κλιματικής αλλαγής το 2019. Α, όχι, είναι το επόμενο αυτό. Αλλά αφού μπορούμε να περάσουμε τώρα σε αυτό, να πάρετε το λόγο, ναι. Στη διάσκεψη των ΟΕΕ για την κλιματική αλλαγή. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να εξηγήσω για ποιο λόγο εγώ απήχα. Απήχα κατά την ψηφοφορία διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που ζητάει είναι πάρα πολύ φιλόδοξη στόχη και καλά κάνει γιατί είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει να στηρίξει τα κρατη για να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλα αέρια. Είναι πολύ φιλόδοξη στόχη πράγματι και το 5% που περιλαμβάνει τις προτάσεις το 2030 είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος αλλά να αυξηθεί πάνω από το 50% χωρίς να γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο, ο, αντίκτυπος των στόχων αυτών είναι κάτι που δεν θεωρώ σκόπιμο να γίνει, γι' αυτό και απήχα. Ζητείται επίσης ε, απαγορεύση παραγωγής ηλεκτρικής ε, ε, χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, αλλά έτσι πολλές χώρες ε, δεν θα μπορέσουν να καταφέρουν του στόχου, γι' αυτό και απήχα, επειδή αυτέ οι παράγραφοι δεν είναι μέσο. Και ο Τζαμπάσκι. Πρόεδρε, εγώ δεν υποστήριξα το ψήφισμα για την ε, επίγουσα κατάσταση του κλίματος, γιατί τα μέτρα που προτείνονται επηρεάζουν την κυριαρχία των κρατών μελών και είναι εις βάρος των συμφερόντων τους. Ε, εγώ διαφωνώ κάθετα με την αύξηση του επίπεδου φιλοδοξίας και της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Συμβολής. Μια τόσο γρήγορη αλλαγή θα ακύρωνε την νομική ασφάλεια και θα κατέληγε σε απρόβλεπτες καταστάσεις για τον κλάδο. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το Brexit, το οποίο θα καταλήξει στην αύξηση των στόχων των άλλων χωρών. Εγώ είμαι από τη Βουλγαρία, μια χώρα που βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης τέτοιοι στόχοι σημαίνουν πως ε, ο κλάδος θα μετεγκατασταθεί σε τρίτες χώρες όπου δεν ισχύουν τέτοια μέτρα. Σας ευχαριστώ. Για το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, θέλετε εσείς ή για αυτό, για, τις για τη διάσκεψη για τις κλιματικές αλλαγές. Μάλιστα. Μάλιστα, έχετε το λόγο τότε κύριε Κέλλη. Εγώ στηρίζω αυτό το ψήφισμα και καλωσορίζω τη φιλόδοξη ατζέντα του Κοινοβουλίου για τις κλιματικές αλλαγές για τα επόμενα πέντε χρόνια με φιλόδοξους στόχους όπως αυτοί εκτέθηκαν και στο Παρίσι. Είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να τιμήσουμε τις επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρξει και διεθνής προσπάθεια για να υπάρξουν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Δεν θα πρέπει να μείνει κανείς πίσω και γι' αυτό και συμφωνώ με τη διάταξη που μιλά για κατάργηση των ορυκτών καυσίνων μέχρι το 2020. Όμως θα πρέπει και να απαγορευτούν μέχρι το 2020 οι κρατικές επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα. Αυτή είναι μια σταδιακή διαδικασία δεν μπορούμε να διακόψουμε απόλυτα τις επιδοτήσεις από τον επόμενο χρόνο, γιατί αυτό θα επηρεάζει και θα επιβάρυνε τις ήδη ευάλωτες οικογένειες. Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να είναι δίκαιη για όλους, αλλά και φιλόδοξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Ο κύριο Τζαμπάσκη. Ευχαριστώ. Καταψήφισα τη συγκεκριμένη πρόταση. Δεν είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει σαν στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι ένα έγγραφο το οποίο ουσιαστικά κάνει προπαγάνδα υπέρ ενός φύλου, μια προπαγάνδα η οποία είναι καταστροφική για τις παραδοσιακές οικογένειες στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Πολλές χώρες είναι κατά αυτής της συμβάσεως όχι ότι είναι υπέρ της βίας, αλλά είναι κατά της συμβάσεως γιατί καταστρέφει ε, τους παραδοσιακούς οικογενειακούς ε, ε, δεσμούς. Δεν μπορούμε να ορίσουμε το φύλλο. Το φύλλο δεν είναι θέμα επιλογής. Το, το φύλλο δεν είναι κοινωνικός παράγων. Το φύλλο είναι αυστηρά βιολογικός παράγων. Σόιντροβα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν θα μπορούσα να στηρίξω ένα ψήφισμα το οποίο να ζητά από όλα τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν άμεσα την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Λουτανία, η Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, ε τους ζητείτε να το κάνουν αμέσως. Νομίζω ότι εδώ πρόκειται για μία μυθοποίηση, μία προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων ότι με την υιοθέτηση της συμβάσεως της Κωνσταντινούπολης θα βρεθούν λύσεις. Η λύση είναι η καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών. Στην Τσεχία έχουμε έναν συγκεκριμένο νόμο Έχουμε μέτρα τα οποία προβλέπονται στον ποινικό μας κώδικα. Έχουμε μέτρα τα οποία προβλέπονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν χρειάζεται να επικυρώσουμε η αδίποτε διεθνή σύμβαση για να κάνουμε αυτό που πρέπει. Αυτή είναι αυστηρή αρμοδιότητα των κρατών μελών και το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να ανακατεύεται. κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ αναγνωρίζοντας ότι η βία εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών δεν αναφέρεται, δεν αποκαλύπτεται. Ε, η οικιακή βία υπήρξαν 8.000 αποδεδογμένες υποθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι στατιστικές δεν πρέπει να έχουν θέση στις κοινωνίες μας και λυπάμαι που η χώρα μου δεν έχει ακόμα υιοθετήσει την συγκεκριμένη διεθνή σύμβαση. Υπάρχουν νομίζω πάρα πολλοί αδύναμοι συμπολίτες μας που χρήζουν προστασίας. Οι κόρες μας, οι αδελφές μας, οι μητέρες μας θέλουν, θέλουν προστασία. Δεν θα πρέπει να πυροβολούν τις γυναίκες όταν σηκώνουν τη φωνή τους, όταν κυκλοφορούν μόνες τους Το 2017 2.700 γυναίκες δολοφονήθηκαν, 80 περίπου χιλιάδες βιάστηκαν και δεκάδες άλλες χιλιάδες υπέστησαν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης bullying ε, είναι κάτι που πρέπει να καταδικάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να περάσουμε τους αυστηρότερους νόμους σε όλα τα επίπεδα. Και το 2019 250 ε, δολοφονίες εις βάρος των γυναικών, το 17 συγγνώμη. Είναι απαράδεκτο που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επικυρώνει ακόμα την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και σύν της άλλης η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει τα χρήματα με τα οποία τροφοδοτεί τις γραμμές καταγγελίας βιασμών και βοήθειας γυναικών. Κύριε Κέλλη, πριν σας δώσω το λόγο, να μας υπενθυμίσω πως ε, για την ε, κατάθεση αιτήματων για τι επεξηγήσει ψήφου. Η προθεσμία λίγη πριν αρχίσει η συνοδοσία. Ε, επομένω μετά δεν γίνεται. Τα έχετε πάντω το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Και στο συγγνώμη που έκανα λάθος και κατέθεσα αργά το αίτημα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ε, σύμβαση, σύμβαση Κωνσταντινούπολης Πολλές έχουν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση ή άλλη φυσική, σωματική κακοποίηση στη ζωή τους και αυτά είναι απαράδεκτα. Πρέπει να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα για να υπάρξει αλλαγή για την κατάσταση και τη ζωή των γυναικών. Αυτή η σύμβαση επικυρώθηκε από την Ιρλανδία νωρί φέτο και επιβάλλει δεσμευτικά πρότυπα κατά τη ε, εμφυλή ε, βία. Η προσχώρηση της Ένωσης είναι κάτι πολύ θετικό, θα βελτιώσει ακόμη τα ε, πράγματα, πιστεύουμε, και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν κάτι το αντίστοιχο άμεσα, δηλαδή να συμπεριλάβουν την, εθνική, ε, την ε, σύμβαση στην εθνική του Και ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Πρόεδρος, πηγαίνω στο επόμενο σημείο που είναι η πρόσφατη ανάγκη τη Ρωσική Ομοσπονδία εναντίον των Λιθανών, δικαστών κτλ. Έχετε το λόγο, κύριε Ολέκα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Οι δράσεις της Ρωσίας, ε, οι ενέργειες μάλλον της Ρωσίας απέναντι σε λιθόνες δικαστές εισαγγελίες και ανακριτές είναι, για, είναι μια ανευπροηγουμένη παρέμβαση στο δικαστικό σύστημα μιας άλλης χώρας. Ε, το κράτος δικαίου πρέπει να είναι αντικείμενο προστασία, όχι μόνο στη Λιθουανία, ε, αλλά παντού. Θα πρέπει να αντιδράσουμε πέραν τις ενέργειες αυτές της Ρωσίας. Με τα ίδια μου τα μάτια είδα τι έγινε στις 30 Ιανουαρίου όταν έβγαλε τεθωρακισμένα στους δρόμους η Σοβιετική Ένωση σε βάρος ε, αθώων ειρηνικών διαδηλωτών και κάποιος από προσπάθησε να τους βοηθήσω. Σήμερα λέμε ξεκάθαρα, κανένας δεν μπορεί να παρεμβαίνει ε, στην ανεξαρτησία ε, του δικαστικού σώματος. Ευχαριστώ. Κύριε Στανόκα. Εγώ καταψήφισα τον εξάρτητο δικαστικό ε, σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν υπάρχει μονοπόλιο. Σε μόνο οι ένοπτες δυνάμεις της Σοβιετικής Ένωση θεωρούνται υπεύθυνοι ε, το Γενάρη του 1991. Θα πρέπει όμως να δούμε ποιοι έχουν ποινικέ ευθύνε, οι δημοσιογράφοι και άλλοι πολιτικοί όπω ο κύριος Παλέτσκης. Λοιπόν, φαίνεται ότι τον Γενάρη του 1991 οι δικοί μας πυροβολούσαν τους συμπολίτε τους. έγιναν διάφορες βαλιστικές έρευνες και φάνηκε ότι υπήρχαν σκοπευτές ελεύθεροι μυστικοί που πυροβολούσαν αμάχους. Ο Αλκίτας μάλιστα κατηγορήθηκε και ότι κατασκόπευε και συνελήφθη. Το τι έγινε λοιπόν το 14 Γενάρη θα πρέπει να διερευνηθεί. Σας ευχαριστώ. Εγώ υποστήριξα αυτό το ψήφισμα Έχω διατελέσει Υπουργό Δικαιοσύνη στην Τσεχική Δημοκρατία και θα πρέπει να στηρίζουμε την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματο σε οποιοδήποτε κράτο μέλο. Δεν, δεν πιστεύω πω είναι θέμα παρερμηνία αυτό που συνέβη ε, αντίθετα από την προηγούμενο ομιλητή. Εδώ έχουμε θέμα ε, του κράτου δικαίου. Για του δικαστέ, οι εισαγγελεί έφτασαν στο συμπέρασμα, ε, εξέφρασαν την, ε, την νομική του γνώμη και κάποια τρίτη χώρα ασκεί διακρίσεις εναντίον τους η Ρωσία. Και γι' αυτό και δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε διαφορετικά τα όσα συνέβησαν το 1991 στη Λουθένια. Πραγματικά θα με ενοχλούσε ένας, ένας δικαστής ή οποιοδήποτε δικαστικός εκπρόσωπος να καταγγέλλεται ή να διώκεται λόγω της νομικής του γνώμης. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, Λιθουανία και γι' αυτό και είναι ζήτημα για όλους μας και για το κράτος δικαίου. Έχουμε τη συνεχιζόμενη ε, διαμάχη για το Airbus και για τις επικρατικές επιδατήσεις ε, στις αεροπορικές εταιρείε που τώρα ε, ξεχύνεται και στις υπόλοιπες εταιρείε. Έχουμε πρώτη απόφαση από τον, από τον ΠΟΕ που πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Τέσσερα κατημέλη έχουν υποδεχθεί. Όλοι αντέδρασαν εντόνως. Η γερμανική, η γαλλική και η ισπανική κυβέρνηση είπαν, και η ευρωπαϊκή κυβέρνηση είπαν ότι θα απαντήσουν με τους, και για τους δικούς τους δασμούς. Όμως ε, η... δεν έχει δοθεί καμία επιδότηση. Οι τόρεις έχουν υπνοτιστεί από τη ΣΥΠΑ συνεχίζονται οι διατλαντικές σχέσεις και το ελεύθερο εμπόριο μετά το Brexit ενάντια σε κάθε απόδειξη. Η ατζέντα του Τραμπ, America First, είναι απειλή για τις βρετανικές θέσεις απασχόλησης και την ευημερία μας, αλλά οι Tories έχουν τυφλωθεί απέναντι σε αυτό. Ο κύριος Τσαμπάσκι. Σας ευχαριστώ. Ε, είναι ε, αυτό το ψήφισμα αφορά ένα σημαντικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν προσπαθεί να ανοίγει την αγορά. Η... Είναι σημαντικό, σημαντική η εξάρτηση από τις αποφάσεις της Washington. Λόγω της ε, διαφορά Airbus-Boeing δεν είναι σωστό να επηρεάζεται ένας ολόκληρος τομέας ε, όπως είναι η βιομηχανία τροφίμων. Ούτε οι καταναλωτέ ούτε οι αγρότες θα πρέπει να είναι όμοιροι σε αυτήν την ε, ε, διαφορά. Θα πρέπει να μειώσουμε και να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας εξηγήσω γιατί ψήφισα υπέρ της πρότασης αυτής. Έχουν υπάρξει ορισμένες ελλείψεις ε, στα αποδεικτικά στοιχεία ε, σχετικά με την Airbus και θα πρέπει να πάρουμε αντίμετρα ε, σε σχέση με τις εισαγωγές από τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά είναι κρίμα που τα γεωργικά προϊόντα είναι αυτά τα οποία θα επιβαρυνθούν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο μεγαλύτερος ε, εισαγωγέας ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να προχωρήσουν σε μια συμφωνία. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε για την περίπτωση της υπόθεσης Boeing γιατί θα καταστραφεί ο αγροτικός τομέας που έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από τις αμερικανικές κυρώσεις. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Φετικό σώμα του ΠΟΕ Κύριε τον Ντάρλινγκ. Υπερψήφισα για πολλούς που υποστηρίζουν το Brexit. Ο ΠΟΕ είναι στην ουσία ο παράδεισος με τον Τραμπ το να κάνει το Μωυσή που θα οδηγήσει τον επιούσιο λαό στην, στους Αγίους Τόπους. Νομίζω ότι έχει πετύχει λόγω της επιμονής του ο Τραμπ εδώ και τρία χρόνια του στόχους του. Και με τις, ε, τα αποτελέσματα των εκλογών δυστυχώς θα αλλοιωθούν από τα ψέματα με τα οποία έχουμε φορτώσει τον Βρετανικό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει η καλύτερη επιλογή για το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λύσει τα θέματα αυτά σε σχέση με τον ΠΟΕ έτσι ώστε ε, να μπορέσουν να επιβιώσουν ε, οι επιχειρήσεις οι εξαγωγικές. Οι τόροι το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν στοιχεία παράδεκτης ρητορική. Τώρα, διαπραγματεύσεις νέας εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ ψήφισα υπέρ, λέει ο κύριος Κέλεχερ, για την εταιρική σχέση με τη ΣΑΚΕ. Ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και νομίζω ότι μια κάποια μορφή ενισχυμένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας θα αποτελέσει ένα ανοιχτό φόρουμ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί και οι χώρες της Αφρικής, του Ειρηνικού και τις καραϊβικές Ανθρώπινα δικαιώματα, κλιματολογικές αλλαγές, υποστήριξη της δημοκρατίας, όλα αυτά είναι θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να δίνει μαθήματα, η Ευρώπη θα πρέπει να ακούει και να μπορέσει να αντιμετωπίσει και αυτή τις δυσκολίες οι οποίες δημιουργούνται από τις δικές μας αποφάσεις και είναι αρνητικές για τις χώρες αυτές. Ας προωθηθεί λοιπόν αυτή η διακοινοβουλευτική συνέλευση, ας αντιμετωπίσουμε τις κλιματολογικές αλλαγές και ας σεβαστούμε το κράτος δικαίου. Τελειώσαμε μέχρι τις 3.